Oké, azt hiszem, hogy elkezdhetjük a munkát. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας, παρακαλώ. Έχει έρθει η ώρα να ξαναρχίσουμε τις εργασίες μας, κυρίες και κύριοι. Και ελπίζω όλοι να φάγατε ένα ωραίο μεσημεριανό, να πιάτε και έναν ωραίο καφέ να συνομιλήσετε και με τους φίλους και γνωστούς και να είστε έτοιμοι για να ξεκινήσουμε το δεύτερο μισό της συνεδριάσεως. Καλωσορίζω την Ντονάτα Βιβάντη, αντιπρόεδρο του EDF. Εγώ προσωπικώς ονομάζομαι Άνταμ Κόσα, ευρωβουλευτής και πρόεδρος της ε, Intergroup για τις ε, αναπηρίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της μεικτής κοινοβουλευτικής ομάδας, της διακοινοβουλευτικής ομάδας μάλλον. Θα προεδρεύσουμε εμείς οι δύο της συνεδριάσεως και σας παρακαλώ τώρα λίγη ησυχία. Nagyon örülök annak, hogy a fogyatékossággal élő emberek Európai Parlamentjén is ugyanúgy. Είναι πολύ μεγάλη λοιπόν η χαρά μου που μπορώ σήμερα να καλωσορίσω στην συνεδρίασή μου εσάς ε, μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασίας όπως έχουμε πάντα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, μπορούμε λοιπόν να εργαστούμε όπως και σε κανονική συνεδρία του Κοινοβουλίου ακούγοντας ο ένας τι έχει να πει ο άλλος και μέσα σε πνεύμα ισότιμης επικοινωνίας. Είναι πολύ σημαντική η εκδήλωση αυτή η σημερινή για μένα και μεγάλη η εμπειρία της συνεργασίας με όλους εσάς, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε προτάσεις για το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και την κρίση ιδιαίτερα. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Αυτό είναι το θέμα της σημερινής μας συνεδρίασης. Ξεκινήσαμε τη δουλειά μας την καλύτερη χρονική στιγμή. Μόλις φτάνει και ο πρώτος μας ομιλητής για το απογευματινό κομμάτι της συναντήσεως. Τον περιμένουμε για να λάβει τη θέση του. Ε, ε, Κυρίες και κύριοι, και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη και αισθάνομαι μεγάλη τιμή που βρίσκομαι εδώ και συμμετέχω στο συντονισμό αυτή της τεράστιας εκδήλωση με τον πρόεδρο τη ομάδα, αφού μοιραστήκαμε μαζί τόσε μάχε και τόσε δεσμεύσει για τα άτομα με αναπηρίε. Χωρίς να χάσω άλλο χρόνο θα ήθελα να σας υπενθυμίσω να τηρείτε τους χρόνους ομιλία κατανοώντας βέβαια ότι το πάθος ε, που σας οδηγεί στο να προσπαθείτε να μιλήσετε όσο γίνεται περισσότερο ε, το κατανοώ, αλλά θα ήθελα να σας ζητήσω να τηρείτε τους χρόνους ε, για να σεβόμαστε όλους τους ομιλητές. Δίνω στο στο λόγο στον πρόεδρο της πολιτικής ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Χάνες Φόμποντα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά. Αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ όλους σας, όλους όσοι οργανώσατε, συνοργανώσατε αυτή την πολύ σημαντική διάσκεψη. Θέλετε να σας τα πω και γερμανικά. Works. the subtitles seem not to work. Α, δεν δουλεύουν οι υπότιτλοι. Να συνεχίσω ή να περιμένουμε λίγο. Yeah, yeah. So we wait. Okay. Να περιμένουμε λίγο. Can I do something? Yes. I would like to make a proposal after. So I think we can proceed. Άρα νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε. Και πάλι, αγαπητοί συνάδελφοι, εκφράζω τη χαρά μου που βλέπω εδώ και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι έλαβαν μέρος στην οργάνωση αυτού του σημαντικού σημαντικής εκδήλωσης διότι χρειάζεται πολύ στράτευση, πολλή προσπάθεια και είναι πολύ σημαντικό το τσέστα εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ένωση ανοιχτή σε όλους, μια ένωση που δίνει ευκαιρίες, που επιτρέπει τη συμμετοχή σε όλους, τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι. Θα έπρεπε να είναι μια ένωση συμμετοχής, συμπερίληψης, ενσωμάτωσης. Το άρθρο 26 του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζει, αναγνωρίζει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, το δικαίωμα ιδιαίτερα να επωφελούνται από μέτρα που εξασφαλίζουν την ανέκτατη τον αυτόνομο βίο τους, κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση και τη συμμετοχή στην ζωή της κοινωνίας τους. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαιώματα ίσα με τους άλλους πολίτες. Για να τα εξασφαλίσουν όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο η μεγάλη τίτλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι και τα κράτη-μέλη, τοπικές κοινωνίες, περιφερειακές αρχές, όλοι απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλοι οφείλουν να σέβονται τις ιδιαίτερες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Αυτός λοιπόν είναι ο ιδιαίτερος στόχος που καλείται να επιτελέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η ευθύνη της εναντί της ε, αξίας και αρχής της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Πρέπει να εξασφαλίζει τις ισότιμες συνθήκες διαβίωσης για οποιονδήποτε, είτε έχει αναπηρία είτε δεν έχει. Σε εποχές όμως κρίσεως και αγαπητοί κυρίες και κύριοι διερχόμαστε το, τρίτο, το πέμπτο έτος ε, κρίσεως οι πιο ευάλωτοι είναι εκείνοι που πλήττονται περισσότερο από τις περικοπές της δαπάνης των κρατών και κυβερνήσεων. Είναι εκείνοι που πλήττονται περισσότερο από τη λιτότητα και ιδιαίτερα τα άτομα με αναπηρία είναι εκείνα τα οποία πληρώνουν τα σπασμένα κατάσταση για την οποία δεν έχουν ε, ευθύνη, δεν είναι υπεύθυνα. Γι' αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό και επιτακτική ανάγκη να προστατευτούν τα άτομα με αναπηρία. Και εγώ στην ομάδα μου, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αγωνιζόμαστε και κατά της αυστηρής λιτότητας, πάνω απ' όλα γιατί βλέπουμε ότι είναι πολύ σημαντικές οι ανάγκες για τα άτομα με αναπηρία για τους πιο αδύναμους στην κοινωνία. Όλες λοιπόν οι συμβάσεις, συμβάσει των Ηνωμένων για τα άτομα με αναπηρία και άλλες, καθιστούν πολύ σημαντικό. Ε, είναι πολύ σημαντικό όχι να τις διαβάζουμε μόνο, αλλά και να τις υλοποιούμε. Έχει έρθει η ώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιήσει την, την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία που έχει κυρώσει και ένας χάρτης ε, για τα δικαιώματα των ΑΜΕΑ, για συμβίωση μέσα στην κοινωνία και για ε, συμμετοχή και ένταξη στο εκπαιδευτικό γίγνεσθε έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ έχουμε να κάνουμε και με, την ε, με μια δημοσιονομική οικονομική κρίση, η οποία μετατρέπεται σε κοινωνική και ανθρωπιστική κρίση. Πρέπει να βρούμε λοιπόν λύσεις για το ε, για το δημόσιο χρέος των κρατών, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να μην λησμονούμε ότι πίσω από αυτά τα νούμερα και τα στατιστικά στοιχεία βρίσκονται άνθρωποι. Άνθρωποι που υποφέρουν από το ζωνάρι που σφίγγουν οι κυβερνήσεις, άνθρωποι που είναι οι πιο ευάλωτοι στις κοινωνίες μας. Κυρίε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ολοκληρώνω αυτή τη σύντομη παρέμβαση με ένα προσωπικό μου βίωμα Είχα την ευθύνη της κυβέρνησης της ε, πόλης της Βιέννης, ιδιαίτερα στον τομέα της χωροταξίας και του σχεδιασμού ε, για αρκετά χρόνια. Είχα επίσης, ήμουν επίσης δραστήριος της μου και στον χώρο της υγείας. Πολλοί λοιπόν οι φίλοι και συνάδελφοι από μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ε, αγωνίζονται για τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες που θα έχουν τα άτομα με αναπηρία. Οι στενοί φίλοι και γνωστοί που για μένα καθιστούν αυτή την εμπειρία όχι μια ευκαιριακή μόνο επαφή, αλλά μια ουσιαστική εμπειρία. Γιατί στη Βιέννη προσπαθήσαμε να βελτιώσουμε ουσιαστικά τις συνθήκες διαβίωσης των ΑΜΕΑ. Ξέρω ότι δεν είναι αρκούν αυτά. Και ομολογώ ότι ποτέ δεν αρκεί ό,τι και να κάνουμε. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει η αρχή αυτή της ενσωμάτωσης της κοινωνίας να ισχύει όχι μόνο σε, ως ένα δίκαιο και ως μια διακήρυξη, αλλά στην πράξη να εφαρμόζεται και να υλοποιείται. Και αυτό γιατί μερικές φορές λεσμονούμε τα πιο σημαντικά θέματα. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι είστε εδώ. Γιατί εσείς μας υπενθυμίζετε ποιες είναι οι ανάγκες σας, ποιες είναι οι δικές μας οι επιτακτικές ανάγκες, να προσφέρουμε βοήθεια σε αυτούς που τη χρειάζονται. Αυτό σημαίνει πολιτική. Η πολιτική είναι να προσφέρουμε βοήθεια σε αυτούς που τη χρειάζονται. Η πολιτική πολλές φορές ή καμιά φορά βοηθούν αυτούς που δεν χρειάζονται πραγματικά βοήθεια. Δεν είναι σωστό αυτό όμως. Πρέπει η βοήθεια να πηγαίνει σε αυτούς που πραγματικά την έχουν ανάγκη και το ζήτημα νομίζω δεν είναι οικονομικό. Γιατί από το σοσιαλιστικό πεδίο και όχι πολύ μακριά. Μαθαίνουμε εδώ από τους Βρετανούς γειτονές ότι η κυβέρνηση, και ας μην είναι σοσιαλιστική, θα πάρει χρήματα από τις μεγάλες επιχειρήσεις για να ε, χορηγήσει επιδόματα και υποστήριξη σε άτομα με αναπηρία. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σαν παράδειγμα. Σα ευχαριστώ εδώ που είστε παρόντες. Ήταν δική μας υποχρέωση να οργανώσουμε και να συμβάλλουμε στη διάσκεψη αυτή και ενώ υποχρέωση όχι τυπική αλλά ένα ουσιαστικό καθήκον. Σας ευχαριστώ θερμά. Ε, Τώρα καλώ τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Φόρου για τα άτομα με αναπηρία για να μας δώσει μια σύντομη απάντηση και ένα σχολιασμό για το όσο ακούσαμε. Thank you. I know we are um, running behind the time and I know also that uh, Mr. President... Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όπως έχω πει και πριν από λίγο καιρό, είναι πολύ σημαντικό οι πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ενώσουν τις δυνάμεις τους προκειμένου τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία να γίνουν πιο ορατά, να προβληθούν περισσότερο και να μπουν πιο ψηλά στην ατζέντα ολόκληρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ολόκληρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχω ενημερώσει κύριε Πρόεδρε, σας το έχω πει, ότι το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ανθρώπων με Αναπηρίες θα απευθύνει επιστολή σε όλες τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις αρχές της επόμενης χρονιάς, προκειμένου να υπάρξει συνάντηση όλων των ηγετών με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για άτομα με αναπηρίες, προκειμένου να ληφθεί υπόψη το ψήφισμα πάνω στο οποίο θα συμφωνήσουμε σήμερα και έτσι να δούμε κατά πόσο μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή. Με τη δικιά σας υποστήριξη, τόσα περιλαμβάνει και με τη στήριξη βέβαια όλων των ευρωπαϊκών οργάνων, αυτά τα οποία συζητήσαμε δηλαδή σήμερα, συζητούμε και στα οποία θα καταλήξουμε. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα το πρωί είπε και το επανέλαβαν κι άλλοι ότι τα άτομα με αναπηρίες πληρώνουν τελικά για μια κρίση για την οποία δεν ευθύνονται. Τα μέτρα λιτότητας αποτελούν κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες σε μια περίοδο όπου η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος, του δημοκρατικού συστήματος στην Ευρώπη αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες, είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον σε αυτό το τομέα, να καλύψουμε το κενό και να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. Σας ευχαριστώ πολύ. Το γνωρίζουμε, το βλέπουμε ότι πιστεύετε στα δικαιώματά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ τον ε, πρόεδρο του ΔΕΦ που προχώρησε σε σχόλια μετά τόσα μας είπε ο πρόεδρος της ομάδας των σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εγώ από την πλευρά μου χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να καλωσορίσω εδώ και την κυρία Βότμαν Κόλ, που είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θέλω να τη ζητήσω, παρακαλώ, να μας μιλήσει και εκείνη για 10 λεπτά για τα θέματα τα οποία συζητάμε εδώ σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ατόμων με Αναπηρίες. Παρακαλώ. Και να απαντήσω λίγο σε αυτά που άκουσα από τον κύριο Βαρδακαστάνη, σε αυτό που είπε εκείνο, ότι ναι, βεβαίω θα φροντίσουμε και συνεργάζομαι και με την κυρία Κόλ για πάρα πολλά θέματα και συμφωνούμε ότι οι επικεφαλεί των πολιτικών ομάδων θα δώσουν συνέχεια στο έτοιμά σα και προσβλέπουμε σε αυτή τη συνάντηση μαζί προκειμένου να συζητήσουμε συγκεκριμένα ποια βήματα, τι μπορούμε να κάνουμε για τα άτομα με αναπηρίες. Σα ευχαριστώ πολύ. Και τώρα βέβαια η κυρία Βόρτμαν Κόλ. Ευχαριστώ πολύ, Χάνες, και ευχαριστώ πολύ και τον συνάδελφο Κόζα. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Η προσβασιμότητα, το θέμα δηλαδή της πρόσβασης, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Είναι κάτι το οποίο αγγίζει έναν στους έξι συμπολίτες μας. Είναι ένα θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε και σήμερα το πρωί εξάλλου. Έχουμε 8 εκατομμύρια Ευρωπαίους, οι οποίοι υποφέρουν από κάποιο είδους αναπηρία. Αν λοιπόν κοιτάξουμε και την τρίτη ηλικία, θα δούμε ότι τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα. Ένας στους τρεις Ευρωπαίους άνω των 75 ετών αντιμετωπίζει α, αναπηρίες οι οποίες περιορίζουν περισσότερο ή λιγότερο τη ζωή του. Λειτουργεί καλά το μικροφωνό μου, ρωτάω μιλήτρια. Ναι, ναι. Έλεγα λοιπόν ότι ένας στους τρεις Ευρωπαίους πάνω των 75 αντιμετωπίζει αναπηρίες που τους περιορίζουν στη ζωή του. Και τα νούμερα αυτά αυξάνουν βέβαια όσο η γύρανση του πληθυσμού προχωράει στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι προφανώς έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής των ατόμων αυτών. Ως κοινωνία λοιπόν εμείς έχουμε την ευθύνη να δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Όμως, είναι πολύ σημαντικό να μπορούν και αυτοί οι πολίτες να προσφέρουν στην κοινωνία. Αλλιώς η απώλεια είναι μεγάλη για όλους, και για εκείνους και για την κοινωνία. Επιτρέψτε μου λοιπόν εδώ να κάνω μια αναλογία. Για 20 χρόνια ο πυρήνας της ευρωπαϊκής ένταξης ήταν η ενιαία αγορά με τις τέσσερις ελευθερίες της. Ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και ατόμων που βασίζεται βέβαια στις αξίες μας που είναι η δικαιοσύνη, ο σεβασμός και η ισότητα, η συμμεταχείριση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τις δικές της οδηγίες και κανονισμούς, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με τις αποφάσεις του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τις δικές του εκθέσεις, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους λόγους της Ευρώπης, όλοι μαζί προσπαθήσαμε να καλύψουμε τα κενά που υπήρχαν στην εσωτερική αγορά. Και εδώ μιλάω για τους φραγμούς που δεν είναι βέβαια δασμολογικοί, για παράδειγμα, η αμοιβή αναγνώριση των διπλωμάτων, η αναγνώριση προδιαγραφών όσον αφορά τα προϊόντα, που κυκλοφορούν στις χώρες μας. Και για να συνεχίσουμε την αναλογία, κάτι άλλο είναι η προσβασιμότητα, που είναι ένα μη δασμολογικό εμπόδιο, το οποίο όμως βρίσκουν μπροστά τους ένα σωρό άνθρωποι στην κοινωνία μας και που δεν μπορούν να υποφεληθούν από την ενία αγορά και δεν μπορούν καν να λειτουργήσουν ικανοποιητικά μέσα στην κοινωνία μας και πλήρως. Αυτό που κάναμε λοιπόν για τα αγαθά, για το κεφάλαιο, για τις υπηρεσίες δεν το κάναμε πλήρως για τους ανθρώπους μας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας σε αυτό το τομέα. Εγώ είμαι πεπισμένη ότι αυτό πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για όλους μας. Εμείς, η οικογένεια του ΕΛΚ, η οικογένεια του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, πιστεύουμε ότι η ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων αποτελεί μία από τις πιο θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μανιφέστο μας, το οποίο υιοθετήσαμε στη Ρουμανία πριν από λίγους μήνες, το ξεκαθαρίζει αυτό και λέει πιο συγκεκριμένα παραθέτω ότι πρέπει συλλογικά να δρώσουμε για να προωθήσουμε την καλά λειτουργούσα ενιαία αγορά που θα προσφέρει θέσεις απασχόλησης, ευκαιρίες και θα προωθήσει υψηλότερα επίπεδα συμμετοχής στην αγορά εργασίας των νέων, όλων των ανθρώπων, των γυναικών, των μεταναστών, των παιδιών τους και των ατόμων με αναπηρίες. Στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουμε συναδέρφους οι οποίοι αντιμετωπίζουν ήδη τέτοια, τέτοιες προκλήσεις αναπηρίας. Και εδώ θέλω να σας πω, ο κύριος Κώσα που είναι εδώ ε, στη Προεδρία, πόσο πολύ μας έχουν βοηθήσει και εκείνος και άλλοι στην καθημερινή μας ζωή έτσι ώστε να μην ξεχνάμε τα προβλήματα αυτά, ώστε να τα λαμβάνουμε υπόψη μας πολύ συγκεκριμένα στις υποθέσεις που εξετάζουμε. Πιστεύουμε ότι έτσι κι αλλιώς τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες πρέπει να αναφέρονται παντού κάθε φορά που έχουμε να κάνουμε με τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 είναι μια στρατηγική η οποία δείχνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θέλουμε να πετύχουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η στρατηγική μας λοιπόν πρέπει να είναι μια στρατηγική στην οποία να ανήκουν όλοι και να μην αποκλείεται κανείς. Και ένας τρόπος είναι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφωνεί με αυτό ομόφωνα. Όσον αφορά τον κύριο Βαρδακαστάνη, όπως είπε, είναι πολύ σημαντικό να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη, αλλά να συνεργαστούμε και με την κοινωνία των πολιτών, με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, μαζί σας, γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε τις προσπάθειές μας να πιάσουν τόπο. Και εμείς ε, στο ψήφισμά μας λέμε ότι θέλουμε περισσότερες πολιτικές για την διαβίου κατάρτιση, θέλουμε ε, περισσότερη συμμετοχή των πολιτών, θέλουμε ε, με μεγαλύτερη ελαστικότητα όσον αφορά την ηλικία συνταξιοδότησης. Και είμαστε ξεκάθαροι στην άποψή μας ότι οι δυνατότητες απασχόλησης για όλους και για τα άτομα με αναπηρίες είναι κάτι που πολύ συχνά αγνοούμε. Η προσβασιμότητα επίσης πρέπει να αποτελέσει κάτι που να θεωρείται απολύτως φυσιολογικό και όχι μόνο στην οικονομία μας αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρη την κοινωνία. Αν πάτε σε ένα ξενοδοχείο οπουδήποτε στην Ευρώπη, δεν αναρωτιέστε αν θα έχει ζεστό ή κρύο νερό ή αν θα έχει μπάνιο στο δωμάτιο. Αυτό είναι κάτι που θεωρείται δεδομένο. Δυστυχώς όμως δεν θεωρείται δεδομένο όλα τα ξενοδοχεία να επιτρέπουν την πρόσβαση στα άτομα με αναπηρίες. Ούτε ισχύει κάτι τέτοιο σε κτίρια γραφείων ή σε σχολεία ή στα πανεπιστήμια ή στα δημόσια κτίρια, στις τάσεις των λεωφορείων, στους συνδρομικούς σταθμούς. Όμως η συνέπεια μιας τέτοιας δυσκολίας σημαίνει κοινωνικό αποκλεισμό. Και αυτό είναι κάτι απαράδεκτο για μας. Εμείς θέλουμε τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να έχουν όλες τις δυνατότητες για προσβασιμότητα. Και γι' αυτό και πιστεύουμε ότι είναι τόσο σημαντικό στις επενδύσεις που κάνουμε για το μέλλον, από την αρχή να έχουμε θέσει τις σωστές βάσεις, τις σωστές προδιαγραφές που να περιλαμβάνουν και την προσβασιμότητα. Εδώ, στο ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουμε να παίξουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει να δημιουργήσουμε ευρωπαϊκές προδιαγραφές, γιατί αλλιώ θα καταλήξουμε σε κατακαιρματισμό της αγοράς, γιατί τα κράτη-μέλη θα εισάγουν τις δικές τους προδιαγραφές, οι οποίες συχνά δεν είναι συμβατές μεταξύ τους. Και το δεύτερο όφελος από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι ότι θα είναι λιγότερο ακριβές οι υπηρεσίες όταν ε, υπάρχει ενία μορφή σε ολόκληρη την Ευρώπη για την προσβασιμότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις οικονομίες. Όλοι έχουμε να αποφεληθούμε από μια ευρωπαϊκή αγορά και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε νέα κέρδη για όλους από τα οποία και εσείς μπορείτε να αποφεληθείτε. Γι' αυτό και πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας είναι η σωστή προσέγγιση. Χρειαζόμαστε πραγματικούς κανόνες και μια κοινή προσέγγιση. Και δεν μπορεί να είναι ένα θέμα που θα τεθεί σε θελοντική βάση, θα είναι προαιρετικό. Όχι, πρέπει να είναι υποχρεωτικό. Και αν πάρουμε τα μαθήματα που πρέπει από τις Ηνωμένες Πολιτείες με την αντίστοιχη πράξη των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1990 για την προσβασιμότητα, τότε βλέπουμε ότι τέτοιες ρυθμίσεις βοηθούν, γιατί επιτρέπουν να υπάρχει κάποια νομική βεβαιότητα για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα επενδύσουν ανάλογα αντί να πηγαίνουμε πίσω και η υπάρχουσα νομοθεσία θα πρέπει να είναι συμβατή με τις αποφάσεις μας αυτές. Αυτό βέβαια ισχύει και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, για 60 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσε έναν χώρο ειρήνης, ευημερίας και ελευθερίας για εκατομμύρια ανθρώπους. Τώρα βρισκόμαστε εν μέσω μιας κρίσης. Όμως, αν κοιτάξουμε τι έχει γίνει στο παρελθόν, αποτελούμε σύμβολο επιτυχίας και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε σήμερα. Έχουμε δείξει ότι οι χώρες μας μπορούν να συνεργαστούν και να συμβιώσουν για το κοινό καλό. Πρέπει να δείξουμε ότι πιστεύουμε ότι το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και σήμερα, ότι μπορούμε την κρίση αυτή να την ξεπεράσουμε και να την κάνουμε το δρόμο προς την ανάπτυξη. Αυτό όμως θα το πετύχουμε μόνο σε συνεργασία μεταξύ μας. Και εδώ δεν πρόκειται μόνο για την απασχόληση, για τα αγαθά, για την οικονομία αυτό το οποίο είναι ακόμα πιο σημαντικό για όλους μας, για το οποίο πήραμε και το βραβείο Νόμπελ στο κάτω-κάτω, είναι το να αναγνωρίζουμε τι έχουμε πετύχει στον τομέα της ελευθερίας και της ειρήνης. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί με τους αυτούς μας, κυρίες και κύριοι. Δεν έχουμε κάνει ακόμα αρκετά προκειμένου η ένταξη και η προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρίες και των ηλικιωμένων να έχει γίνει πραγματικότητα. Ελπίζω ότι τα βήματα που λαμβάνουμε σήμερα είναι τα πρώτα βήματα, αλλά αποφασιστική σημασίας προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ευρώπη πρέπει να γίνει ε, ηγετικό στοιχείο στον αγώνα αυτό. Δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα, αλλά μπορείτε να βασιστείτε στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για να τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστούμε πολύ κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας και ευχαριστούμε που τηρήσατε και το χρόνο ομιλίας. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του EDF, του Ευρωπαϊκού Φόρουμ. I and we have listened Ακούσαμε μόλις ε, μια πολύ ακριβή παρουσίαση του πώ ακριβώ θα έπρεπε να είναι, τι εικόνα έπρεπε να έχει η προσβασιμότητα. Από... Μας είπε η Αντιπρόεδρος ε, πως ε, θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική η ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας και συμφωνήσαμε ήδη ότι θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Μπροστά μας, το 2013, Έχουμε σημαντικά ζητήματα να επιλύσουμε και νέα ζητήματα για τα οποία θα πρέπει να αγωνιστούμε. Πρέπει να ολοκληρώσουμε του ε, διάφορους κανονισμούς, ε, την εξωτερική βοήθεια, όπου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται ε, τα δικαιώματα όπως προβλέπονται από τα Ηνωμένα Έθνη. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα χρειαστεί να συζητήσει την νομοθεσία η οποία προτάθηκε στις 3 Δεκεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο και θα προσπαθήσουμε να ε, λάβουμε την υποστήριξη του Κοινοβουλίου, να είναι αυτή η υποστήριξη πιο ευρεία, πιο αποτελεσματική, να καλύπτονται όλες, όλοι οι ιστότοποι, να προσφέρονται περισσότερες υπηρεσίες στο κοινό. Φυσικά η ευρωπαϊκή πράξη προσβασιμότητας θα προταθεί στα μέσα του έτους. Έχουμε λοιπόν πολλά να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και θα πούμε και σας αυτό που είπαμε στον προηγούμενο μιλητή. Θα στείλουμε μια επιστολή σε όλους τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων στο Κοινοβούλιο ώστε να συναντηθούμε με το Ευρωπαϊκό Κίνημα για Άτομα με Αναπηρίες και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τα λόγια πράξης σε αυτές τις εποχές ε, ταραχών, ταραγμένες εποχές τις οποίες ζούμε. Είναι σημαντικό να ακούμε φωνές όπως η δική σας που να στηρίζουν το έργο μας και να τονίζουν τις ανάγκες ε, που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίε και οι οικογένειε του σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ. Ehm. Ευχαριστούμε. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Ίνεξ Κριστίνα Τσούμπερ, Αντιπρόεδρο της Επιτροπής ε, Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω ισπανικά, γιατί πορτογαλικά δεν έχουμε, λέει μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα μου, λέει Είμαι πορτογαλέζα, οπότε είναι και αυτό κάποιο είδου διάκριση, τότε δεν μπορώ να μιλήσω τη γλώσσα μου, λέει η ομιλήτρια. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ σήμερα. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση αυτή. Και θέλω να σας μεταφέρω μερικά πράγματα, τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με την ε, δουλειά μας, αλλά έχουν να κάνουν και με τη χώρα από την οποία προέρχομαι. Γιατί μιλάμε για την κρίση εδώ. Η χώρα μου, η Πορτογαλία, βρίσκεται εν μέσω κρίσης ε, βεβαίως πολύ σοβαρή κρίσης και τις συνέπειες τις νιώθουν όλοι όλες οι πλευρές της κοινωνίας, αλλά εννοείται τα άτομα με αναπηρίας ακόμα περισσότερο. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι πριν από ένα χρόνο στην Επιτροπή, την κοινοβουλευτική όπου συμμετέχω, δηλαδή κοινωνικών υποθέσεων, εγκρίναμε μία έκθεση του συναδέρφου Άνταμ Κόσα ακριβώς, που είχε να κάνει με την σημασία που έχουν οι πολιτικές λιτότητας και πώς πλήττουν τα άτομα με αναπηρίες. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όμως, εγώ είμαι κάπως πιο απεσιόδοξη. Γιατί, γιατί πιστεύω ότι στην πραγματικότητα οι πολιτικές λιτότητας επηρεάζουν πάρα πολύ τα άτομα με αναπηρίες. Και γιατί? Γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως είπαμε, πλήττουν ε, όλους τους τομείς. Λοιπόν, αν πλήττουν τους εργαζόμενους, επλήττουν και τους εργαζόμενους με αναπηρίες. Αν υπάρχει ανεργία στην κοινωνία γενικά, ε, υπάρχουν ακόμα περισσότερες δυσκολίες για δουλειά για τα άτομα με αναπηρίες. Αν υπάρχουν μισθοί που μειώνονται, είναι πιο χαμηλοί, εμειώνονται και για τα άτομα με αναπηρίες. Δηλαδή, αυτά έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μεμονωμένες οι περιπτώσεις των αναπήρων. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι υπάρχει ένα κενό, μεγάλο κενό, ένα χάσμα ανάμεσα στα επίσημα όργανα, όπως είναι για παράδειγμα η Σύμβαση αυτή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και της πραγματικότητας. Χάσμα ανάμεσα στα δύο. Η κοινωνική πραγματικότητα βρίσκεται μακριά. Και αυτό το χάσμα βαθαίνει όλο και πιο πολύ. Και γιατί. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη οπισθοχώρηση αν εμείς αντικαθιστούμε την ιδέα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, βασικά δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζονται από το κράτος, γιατί είναι δικαιώματα, αν λοιπόν αντικαταστήσουμε αυτά από μία φιλοσοφία φιλανθρωπίας, κοινωνικής επιδότησης. Γιατί αυτό πλήττει την αξιοπρέπεια των ατόμων με αναπηρίες. Τώρα για να μιλήσουμε λίγο και για την θεωρία αυτή πιο πολύ. Αν εμβαθύνουμε λιγάκι στα θέματα έλλειψης κοινωνικής δικαιοσύνης, όταν υπάρχει μια πιστοχώρηση των κοινωνικών δικαιωμάτων και των εργασιακών ε, δικαιωμάτων, η κοινωνία δεν θα μπορέσει ποτέ να πετύχει την ε, συμμετοχή όλων στην κοινωνία. Όλα αυτά τα λέω γιατί ξέρω τι συμβαίνει στη χώρα μου και πώς έχουν πληγεί τα δικαιώματα των ατόμων ε, με αναπηρία στην ε, Πορτογαλία. Με από τις περικοπές στον προϋπολογισμό έχουν επηρεαστεί πολύ τα επίπεδα προστασίας των ατόμων με αναπηρίες. γίνονται περικοπές στο κοινωνικό επίπεδο πολύ μεγάλες για τα άτομα αυτά. Για παράδειγμα, οι συντάξεις για τα άτομα με αναπηρίες. μετά από εργασιακά ατυχήματα. Υπάρχει ένα πάγωμα. Οι περισσότεροι από αυτούς παίρναν 407 ευρώ και τώρα παίρνουν τα ίδια παρόλο που υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Η αύξηση στη φορολογία. Και αυτή πλήττει τα άτομα με αναπηρίες. Πρέπει να πληρώνουν περισσότερους φόρους. Οι περικοπές σε όλες τις κοινωνικές παροχές τους πλήττει επίσης. Και όχι μόνο αυτό. Αν μιλάμε για περικοπές δημοσίων δαπανών, πρέπει να μιλήσουμε για περικοπές σε στήριξη επιστημονικών έργων, λογοτεχνικών έργων, πολιτιστικών αγαθών, περικοπές στα χρήματα που δίνονται για την νοηματική γλώσσα για την προσαρμογή των κτηρίων ώστε να υπάρχει πρόσβαση εύκολη των ατόμων με αναπηρίες κλπ. Δηλαδή, δεν μπορούμε το θέμα αυτό της ένταξης των ατόμων με αναπηρίες να το δούμε μεμονωμένα. Γιατί αν υπάρξουν στις κοινωνικές πολιτικές και γενικά στις πολιτικές μιας χώρας περικοπές, απευθείας πλήττονται και τα άτομα με αναπηρίες. Άρα δεν θα είμαστε σε θέση να τηρήσουμε τα τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών. Και ζητώ συγγνώμη που τα λέω έτσι ομά, αλλά βλέπετε, εγώ φοβάμαι ότι η σύμβαση με την πραγματικότητα βρίσκονται έτη φωτός μεταξύ τους σε απόσταση. Φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Στην εργασία πρέπει να υπάρξουν προγράμματα ένταξης. Για να βοηθήσουμε τα άτομα με αναπηρίες να έχουν πρόσβαση στην απασχόληση. Αν δεν αλλάξει λοιπόν ριζικά η βάση των πολιτικών, τα διάφορα δικαιώματα τα οποία διασφαλίζει η σύμβαση δεν θα τηρούνται. Αντίθετα θα πηγαίνουμε πίσω και δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τίποτα αν δεν αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο κάνουμε πολιτική γενικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Αντιπρόεδρε. Δίνω τώρα το λόγο στον Άλλαν Φόγο, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα άτομα με αναπηρία. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, από σήμερα το πρωί δεν έχουμε σταματήσει να διαπιστώνουμε ότι η οικονομική κρίση σιγά σιγά μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε κρίση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, κυρώσει την ε, συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία και τι πρέπει να κάνουμε για να εφαρμόσουμε αυτή τη συνθήκη στην πραγματικότητα. Για να αντιμετωπίσουμε την κρίση πρέπει να προβληματιστούμε και να υλοποιήσουμε καλύτερα, να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τους χρηματοοικονομικούς πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρώτα απ' όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να υιοθετήσουν ένα ισχυρό πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει τι κοινωνικέ επενδύσει, ώστε να βγούμε από την σημερινή οικονομική και κοινωνική κρίση, να κατανέμει επαρκές ποσό των διαρθρωτικών ταμείων, και να κάνει προσβάσιμες στις διατυπώσεις για την πρόσβαση σε αυτά τα διορθωτικά ταμεία. Να βεβαιωθεί ότι τα μελλοντικά διορθωτικά ταμεία θα χρηματοδοτήσουν την προσβασιμότητα και την συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και να υποστηρίξουν τα έργα δικτύων υποδομών με προσβασιμότητα. Την ανάπτυξη συγκεκριμένων δικτών ε, αναπηρίες, ε, συλλογή πληροφοριών, ώστε να γνωρίζουμε καλύτερα τις ε, κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται από την κρίση και υλοποίηση εξατομικευμένων λύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί να αναπτύξει ένα κοινωνικό επενδυτικό πρόγραμμα βασισμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις μη διακρίσεις ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ως μέλος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό το πρόγραμμα, το μακροπρόθεσμο θα πρέπει να επικεντρωθεί σε κοινωνικές πολιτικές που θα καταλήξουν σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμού. όλο και περισσότερο. Και με μεγαλύτερη ευημερία πρέπει να υποστηρίξει την έννοια της ελάχιστης κοινωνικής προστασίας όπως έχει εκμονηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Εργασίας και να ορίσει τις βασικές υποχρεώσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων περιλαμβάνοντας πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες όπως νερό, υγεία, υπηρεσίες υγεία, ε, μεταφορές, εκπαίδευση, όλα αυτά τα οποία είναι απαραίτητα για τους αναπήρους οι οποίοι είναι όλο και περισσότερο εκτεθειμένοι στην ένδυα καθώς και ένα ελάχιστο εισόδημα και πρόσβαση σε βασικές ε, ε, υπηρεσίες αρρωγής όπως υπηρεσίες υγείας. Θα πρέπει αυτό να αποτελέσει τη βασική αρχή για την προστασία των ατόμων με αναπηρία. Αγαπητοί φίλοι, Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί οργανισμοί, έχουμε υποχρέωση να υπερασπιστούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα βάσει της συνθήκης των Ηνωμένων για την προστασία των ατόμων με αναπηρία. Όσοι είστε υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων, φέρετε μεγάλη ευθύνη το να υλοποιήσετε αυτή την συνθήκη και να αποφύγετε αυτή την κρίση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Köszönöm szépen Σας ευχαριστούμε πολύ. Το πρώτο τμήμα λοιπόν της απογευματινής μας συνεδρίασης ολοκληρώνεται και προχωρούμε για να ακούσουμε τις ε, επεμβάσεις επί της ουσίας από τους συναδέλφους αλλά θα ήθελα προηγουμένως να προσθέσω εγώ κάποια σημεία προσπαθώντας να σκιαγραφίσω τον τρόπο με τον οποίο Κοινοβούλιο και εγώ και άλλοι προσπαθούμε να προβάλλουμε τα ζητήματα των ατόμων με αναπηρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τις εξελίξεις έτσι ώστε η νομοθεσία να έχει να λαμβάνει πραγματικά υπόψη τα ζητήματα των ΑΜΕΑ. Εγώ προσωπικώς είμαι ΑΜΕΑ. Καθημερινά αντιμετωπίζω τις δυσκολίες, τα εμπόδια που έχουν όλα τα άτομα με αναπηρία. Και πιστεύω ότι εάν θέλει κανείς μπορεί πράγματι να συμβάλλει στο να εξασφαλιστούν, να παραχ ληφθούν καλά νομοθετήματα, νομοθετήματα τα οποία θα δυσφαλίζουν καλέ συνθήκε. για τα νέα. Θα δώσω λόγο τώρα στον κύριο Τόισεν, διευθυντή του EDF. Ε, Αναμένοντα τον κύριο Έρικ Όλσεν, μέλο τη εκτελεστική επιτροπή του EDF ε, και εγώ ω αντιπρόεδρο του EDF θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια για αυτό το κρίσιμο επιχείρημα που είναι ο τρόπος, ο οδός εξόδου από την κρίση. Τι σημαίνει και πώς μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς ε, να συνεχίζουμε αυτή την παραβίαση, την καταπάτηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία όπως έχει γίνει μέχρι σήμερα και όπως αναγνωρίζεται στη συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών. Είναι σαφές ότι ο οδός εξόδου από την κρίση θα απαιτήσει αλλαγή νοοτροπίας και στάσεις προς τα άτομα με αναπηρίες ώστε να αξιοποιηθεί ο πλούτος που για παράδειγμα οι νέοι και τα παιδιά με αναπηρίες διαθέτουν και αποτελούν για ολόκληρη την κοινωνία μας. Απαιτεί όμως και συγκεκριμένες επενδύσεις. Απαιτεί επίσης ε, και προσπάθειες ώστε η εξάρτηση και η περαιτέρω αναπηρία που δημιουργείται, που προκαλείται όταν δεν υπάρχει ανταπόκριση στις απαιτήσει στήριξης του κάθε ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ιδιαίτερες απαιτήσει υποστήριξης, θα έχει συνέπειες και πάλι στις μελλοντικές γενιές. Συνεπώς, η οδός εξόδου από την κρίση πρέπει υποχρεωτικά να διέλθει από τη συμμετοχή όλων των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία μας. Πρέπει επίσης να βασιστεί και στη συμμετοχή των ατόμων ε, με αναπηρία στην, ε, στη χάραξη πολιτικών δράσεων ώστε κανείς να μην ξεχαστεί, να μην εγκαταλειφθεί στο μέλλον. Δεν θα... Χωρίς άλλο χάσιμο χρόνο λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Την Ολομέλεια, πρώτος ε, ομιλητής στη λίστα είναι ο κύριος Νικόλσεν ο οποίος ωστόσο δεν βρίσκεται ακόμη στην αίθουσα θα μας συγχωρέσετε αν κάνουμε κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα κάποια άτομα πρέπει να φύγουν πιο γρήγορα δίνω λοιπόν το λόγο στον Πύρκο Μαλαμάκη ε, γραμματέα της Φιλανδικής Ομοσπονδίας για άτομα με αναπηρία και θα ζητήσω να ετοιμαστεί η Τσεκλεντίν Κόμματς Άβετς της Ουγγρικής Ομοσπονδίας για άτομα με αναπηρία. Ε, ε, θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω όταν πρόκειται να μιλήσετε να σηκώνετε το χέρι ώστε να μπορέσει να σας βρει ο κάμεραμαν. On behalf of the εκ μέρου του Φιλανδικού Φόρουμ Αναπηριών θα ήθελα να απαντήσω στο ερώτημα του πώς μπορούμε να διαφύγουμε από την κρίση. Σήμερα το πρωί ξεκινήσαμε μιλώντας για την, για την ανάγκη για μια νέα και σαφέστερη νομοθεσία για τις αναπηρίες. και υπογραμμίστηκε ότι μπορεί η πίεση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον προχωρήσει αυτή σε νομοθεσία, θα, αντανα... θα έχει την ανάκριση και στην εθνική νομοθεσία. Έτσι λοιπόν ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας θα υλοποιήσει τις ελπίδες που όλοι τρέφουμε. Επίση, θα θέλαμε για ένα συγκεκριμένο σημείο και, εκ της εθνικής, και από την εθνική μας ακριβώς εμπειρία να αναφερθούμε στο ζήτημα τη υλοποίηση, που είναι ένα από τα κύρια μέσα για να ξεφύγουμε από την κρίση διότι η υλοποίηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών είναι η καλύτερη βάση για τη δημιουργία μιας Ευρώπης όπου όλα τα αμαία είναι χρήσιμα στις κοινωνίες τους, εντάσσονται στην, ε, στον επαγγελματικό βίο, στην εκπαίδευση, στον εκπαιδευτικό βίο, ως χρήσιμα άτομα για τις κοινωνίες τους. Και έτσι μπορούμε απλώ να υπογραμμίσουμε την ε, σημασία των, και τις υποσχέσεις της Συμβάσεως των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να πω ότι δυστυχώς η χώρα μου ακόμα δεν έχει ολοκληρώσει την κύρωση. Ελπίζουμε ότι θα το πράξει το χειτερό δυνατό. Και μια τελική παρατήρηση για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία κατά των διακρίσεων. Το κίνημα των ατόμων με αναπηρία επέτυχε να βελτιώσει μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο την κατάσταση των διακρίσεων εις βάρος των ΑΜΕΑ. Επιδιώκουμε λοιπόν να διευδυνθεί αυτό το φυστάμενο πλαίσιο. Ένα πλαίσιο που χρειάζεται, ένα πλαίσιο που θα θέλαμε να δούμε να επανέρχεται, ιδιαίτερα εγώ και άλλα άτομα με αναπηρία σε χώρες όπως η Φιλανδία, όπου έχει σημαντικά υποβαθμιστεί η προστασία με επιχείρημα την κρίση. Μα η απάντηση στην κρίση νομίζω είναι ακριβώς αυτή την οποία δώσαμε με την ε, σύμβαση. Τίποτα που να μας αφορά χωρίς εμάς. Τίποτα για μας χωρίς εμάς. Ευχαριστώ. Κόβας και παρακαλώ τον κύριο Χριστονάστα να ετοιμάζεται. Θα είναι ο δεύτερος ομιλητή. Παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σημειώνουμε, Πρόεδρε, θετικές ραστηριακές αλλαγές ως προς την νομοθεσία που υιοθετείται, μια νομοθεσία η οποία βελτιώνει την ισότητα ευκαιριών. Πολλά ήταν τα προβλήματα που είχαμε Εσφαλμένες κυβερνητικές πολιτικές επιδίνωσαν την κατάσταση. Είδαμε ακόμη και οπισθοδρόμηση. Και έτσι άτομα με αναπηρία μετατρέπονται στους μεγάλους χαμένους της οικονομικής κρίσης καθώς ε, περικόπτονται οι προϋπολογισμοί και αντίστοιχα οι υπηρεσίες, η προστασία, τα επιδόματα που προσφέρονται στους, στα άτομα με αναπηρίες, που προβλέπονται για τα άτομα με αναπηρίες. Περικόπτονται τα σχετικά ποσά στον προπολογισμό όταν είχαν προβλεφθεί ή όπου είχαν προβλεφθεί για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των ατόμων με αναπηρία, αλλά αυτέ οι περικοπέ δεν έχουν βοηθήσει σε τίποτα την οικονομική κατάσταση. Παραμένει χαμηλή η ανεργία, παραμένουν οι μισθοί και τα εισοδήματα σε πολύ πολύ χαμηλό επίπεδο. Και η απασχόληση σε διάρκεια χαμηλότερη των τριών μηνών. Έτσι λοιπόν πρέπει πιστεύουμε να δώσουμε καινοτόμες λύσεις με στόχους, με αποκατάσταση, με απασχόληση, με άλλες πολιτικές, γιατί εδώ δεν μιλούμε για, για ελεημοσύνη, δεν μιλούμε για φιλανθρωπία για τα αμαία. Εδώ μιλούμε για επένδυση που αποδίδει ουσιαστικά και γι' αυτό θέλουμε τα ΑΜΕΑ να έχουν θέσει εργασίας στην ανοιχτή αγορά. Θέλουμε πολιτικές οι οποίες θα βοηθούν τα άτομα με αναπηρία, γιατί αυτό είναι το συμφέρον των πάντων. Και πιστεύω ότι πια πρέπει τα λόγια να τα ακολουθήσουν έργα. Με απτές πρωτοβουλίες, προς το συμφέρον όλων μας. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστούμε. Το λόγο έχει τώρα ο Χρήστος Νάστας του Συμβουλίου για τα άτομα με αναπηρία τη Ελλάδα, Γενικός Γραμματέας και θα ζητήσω από τον Βακλαβ Κράζα του Συμβουλίου για τα άτομα με αναπηρία της Τσεχικής Δημοκρατίας να προετοιμαστεί για την επόμενη ομιλία του. Χρήστος Νάστας. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του EDF, κύριε Ευρωβουλευτά, κυρίες και κύριοι, Η χώρα μου η Ελλάδα βιώνει σήμερα τη βαθύτερη οικονομική κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τον πολίτη αναπηρία και χρόνια πάθηση που θα έπρεπε να είναι το κεντρικό πρόσωπο των εφαρμοζόμενων πολιτικών κοινωνικής προστασίας, ειδικά σε μια χώρα με αποκλεισμένα μέσα στο μεγάλο νησιωτικό σύμπλεγμά της, οι πολιτικοί οργανισμοί και τα στελέχη τους τον εγκαταλείπουν στην τύχη τους, έχοντας μετατραπεί σε δικαστικούς επιμελητές επίδοσης των αποφάσεων της Τρόικα. Και εκτιμένα με αγώνες του αναπηρικού κινήματος την τελευταία 25 ετία, καταραίουν ως χάρτινος πύργος. Προγράμματα από ασυλοποίησης, επιδόματα, δομές ημερήσιας φροντίδας και αποκατάστασης κλείνουν τον κύκλο τους η επιστροφή σε ιδρύματα που η κρίση έχει μετατρέψει σε χώρους αφιλόξενους τρομάζει, γυρίζοντας τη σκέψη σε κολαστήρια τύπου Λέρου. Το ερώτημα που βγαίνει σαν κραυγή αγωνίας από το στόμα των αναπήρων πολιτών είναι ένα. Πού μας οδηγούν, σε ποιο είδος κοινωνικής ευθανασίας. Μήπως φτάσουμε στο σημείο να δούμε στρατιές αστέγων και των αναπήρων να κλείνουν τον κύκλο τους στους δρόμους. Κυρίες και κύριοι, προστασία κάτω από αυτές τις αφιελτικές συνθήκες παρέχουν δύο μόνο εργαλεία που είναι τα ακόλουθα. Πρώτον, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ και το προαιρετικό πρωτόκολλο που έχει κυρώσει η χώρα μου όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, η προσφυγή στα όργανα και τις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή όλων των μέτρων και των πολιτικών που έχει θεσπίσει για τα άτομα με αναπηρία. Η, αξιοποίηση αυτών των σημαντικών εργαλείων μπορεί να φέρει ανατροπές όταν οι στοχευμένες κινήσεις εκπορεύονται από το Εθνικό Αναπηρικό Κίνημα που διαθέτει τεχνογνωσία, ευρωπαϊκή και διεθνή εμπειρία μέσα από τη συμμετοχή του στο European Forum και στην Άιντα. Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας, ανάπηροι και γονείς ατόμων με αναπηρία, σας καλούμε να στηρίξετε τον αγώνα μας που είναι και δικό σας, γιατί η οικονομική κρίση δεν έχει σύνορα. Απλώνεται σαν τοξικό νέφος πάνω από ολόκληρη την Ευρώπη. Η ενιαία αντίστασή μας θα ανατρέψει τις πολιτικές εκείνων που θέλουν να σβήσουν από την Ευρώπη του πολιτισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το κοινωνικό κράτος. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Δίνω τώρα το λόγο στον Βάκλαβ Κράζα, του Εθνικού Συμβουλίου για τα άτομα με αναπηρία της Δημοκρατίας της Τσεχίας και θα ζητήσω να ετοιμαστεί ο Κρίσταλ Πράντο του Γαλλικού Εθνικού Συμβουλίου για τα άτομα με αναπηρία. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Απόψε έχουμε την έγκριση του ψηφίσματος για την κρίση για τα επόμενα δέκα χρόνια και θα ήθελα και να υπογραμμίσω εκείνο το τμήμα του ψηφίσματος που μιλάει όχι για τη βελτίωση της κατάστασης για τα άτομα με αναπηρία αλλά να πω επίσης ότι όσο και αν δεν είναι τόσο κακή η οικονομική κατάσταση στην Τσεχία η κυβέρνησή μας αποφάσισε να προωθήσει μια πολιτική αυστηρής λιτότητας χάνονται κοινωνικές μεταφορές για τα άτομα με αναπηρία, για τις οικογένειες με μικρά παιδιά, για τους πιο αδύναμους και τα χρήματα που χορηγούνταν, τα επιδόματα και όλα αυτά που χορηγούνταν σε άτομα με αναπηρία έχουν περικοπεί κατά 50%. Έτσι, πολλές είναι οι οικογένειες πλέον που δεν μπορούν να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους. Ε, αντίστοιχα μέτρα περιορισμού βλέπουμε και στο χώρο της απασχόλησης ιδιαίτερα στον ε, ΑΜΕΑ και πιστεύω ότι ε, για να υλοποιηθούν, για να εφαρμοστούν τα άρθρα της Διεθνούς Σύμβασης πρέπει εξάπαντος να έχουμε κοινέ προδιαγραφές, κοινέ αρχές μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προσφέρεται η υποστήριξη στα άτομα με αναπηρία. Δεν είναι δυνατόν ε, για τα κράτη-μέλη να συμφωνήσουν να αποκλείσουν τα άτομα με αναπηρία από την καταβολή δύο-δύο επί παραδείγματι. Νομίζουμε χρειάζεται σαφείς προδιαγραφές, απλές προδιαγραφές για όλα τα άτομα με αναπηρία απλές αρχές που αποτελούν το μόνον τρόπο να υλοποιηθεί η Σύμβαση των Η κρίση που διερχόμαστε πολλές φορές αξιοποιείται από ορισμένου για την αποδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους. Εμείς πρέπει να ταχθούμε σε αυτό και πρέπει ενωμένοι να το καταπολεμήσουμε. Σας ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστώ Βάκλαβ. Δίνω τώρα το λόγο στον εκπρόσωπο του Γαλλικού Εθνικού Συμβουλίου και ζητώ να ετοιμαστεί ο Λουίς Άιγο Κουέρβας, Ισπανός. Καλημέρα. Ποια στρατηγική λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε για να βγούμε από την κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ο τόπο οικοδόμηση της κοινή μας ζωή στην Ευρώπη ένα παγκόσμιο και δημοκρατικό οικοδόμημα. Η κρίση απειλεί όλα αυτά. Δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κρίση παρακατανοώντας καλύτερα ο ένας τον άλλο. Τα άτομα με διανοητικές δυσκολίες ε, έχουν δημιουργήσει ένα εργαλείο το οποίο θα μας βοηθήσει να βγούμε από την κρίση το οποίο θα επιτρέπει σε κάθε γλώσσα της Ένωσης ε, να ε, ε, απλοποιεί τις δύσκολες έννοιες πληροφορικής και κειμένων. Η ομιλία του Γάλλου Πρωθυπουργού απλοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο ώστε να επιτρέψει σε περισσότερους Ευρωπαίους να καταλάβουν, να οικειοποιηθούν καλύτερα περισσότερες γλώσσες της Ένωσης να διευκολυνθούν έτσι οι πολιτιστικές ανταλλαγές και η δημιουργία μεταξύ όλων και να ε, συμμετέχουν όσοι συμμετέχουν στη δημοκρατία μας. Αυτό ε, το μέσο θα βοηθήσει τους πάντες και θα βοηθήσει τα άτομα αναπηρίας να βγουν από τη λογική αρρωγής και να συμμετέχουν στη δημοκρατία ως πολίτες ε, ολοκληρωμένοι. Αυτό θα αποτελέσει τον ορίζοντά μας για να βγούμε από την κρίση. Πώς θα διευκολύνουμε την ανάπτυξη εντός της Ένωσης σε όλα τα μέσα. Αυτή είναι η ερώτηση την οποία θέτω εγώ στο Κοινοβούλιο μας. Ε. Ευχαριστούμε. Να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα τη σύνοψη και την ακρίβεια του επιχειρηματός σας. Τώρα δίνω το λόγο στον Χωσ Λουίς και θα ζητήσω να ετοιμαστεί η Μαρία Γιωχάνσον τη Σουηδική ομοσπονδία για τα άτομα με αναπηρίες. Ε, Καλησπέρα σε όλους σας. Εδώ και 30 χρόνια στην Ισπανία βάλαμε ένα στίχημα προκειμένου να συμμετέχουν στην εκπαίδευση όλα τα άτομα με αναπορίες και βάλαμε σχετικά πράγματα στην νομοθεσία ώστε να στηρίζονται οι μαθητές όποια αναπηρία και αν είχε ο καθένας. Επίσης προβλέπεται η βοήθεια στις οικογένειες, ειδικοί δάσκαλοι, καθηγητές και πρόσβαση στα εκπαιδευτικά κέντρα. Και αυτά είναι κάποια στοιχεία τα οποία βοήθησαν βέβαια στη συμμετοχή όλων στην εκπαίδευση. 3,3% είναι οι μαθητές της υποχρεωτικής ε, εκπαίδευσης που εκπαιδεύονται σε ειδικά κέντρα. Ιδιαίτερα δώσαμε σημασία στην περίπτωση των κοφών μαθητών και στις οικογένειές τους. Από ό,τι φαίνεται, αν δοθεί η βοήθεια που χρειάζεται για να συμμετέχουν όλοι αυτοί οι μαθητές στην εκπαίδευση, τα αποτελέσματα είναι τα καλύτερα δυνατόν. Οι περισσότεροι από τους μαθητές αυτούς συμμετέχουν στην εκπαίδευση στο επίπεδο ακριβώς που ταιριάζει με την ηλικία τους. Το 90% των παιδιών και των ε, ε, των ατόμων που βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση, τα παιδιά χρησιμοποιούν την ειδική γλώσσα. Επίσης, τους βοηθάμε για να διαλέξουν και το κατάλληλο σχολείο. Παρ' όλα αυτά, πολλά πρέπει να λυθούν ακόμα. Με την κρίση που έχουμε, γίνεται εξορθολογισμός βέβαια των δαπανών, οπότε πλήττονται και τα άτομα αυτά που σας ανέφερα. Για παράδειγμα, υπάρχουν λιγότεροι ειδικοί στην ε, βοήθεια έκφρασης των παιδιών που έχουν δυσκολία να εκφραστούν. Εγώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι κάτι οριζόντιο και είναι κάτι το οποίο βοηθάει στη συνέχεια την πρόσβαση στην απασχόληση και έχει να κάνει με τα βασικά δικαιώματα των πολιτών. Συνεπώς, οι άνθρωποι με αναπηρίες, αντί να γίνονται άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν χρήματα, γίνονται άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν στην κοινωνία εφόσον τους δώσουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην κοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή σας την παρέμβαση. Πριν δώσω το λόγο στη Μαρία Γιωχάνσον της Σουηδικής ε, Ομοσπονδίας για τα άτομα με αναπηρία. Θα ήθελα να χαιρετήσω όλους σας. Ζήτω συγγνώμη που πρέπει να εγκαταλείψω αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα σύνοδο λόγω τις ώρες αναχώρησης της πτήσης μου και αφήνω τη διεύθυνση της ε, συνόδου στον πρόεδρο της ομάδας, Ανταμ Κόζα, Μαρία Γιωχάνσον, λοιπόν για τη Σουηδική Ομοσπονδία για τα άτομα με αναπηρία. Ευχαριστούμε πολύ. Οι προσβάσιμες υπηρεσίες είναι αναγκαίες. Πρώτα απ' όλα, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε πλήρως τα ανθρώπινα και πολιτικά μας δικαιώματα. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους, ξεκινούν από διαφορετικά σημεία αφετηρίες, αλλά πρέπει να τα δούμε όλα από τη σωστή προοπτική. Τίθεται θέμα δημοκρατίας και αποτελεί προϋπόθεση για βιώσιμη, δίκαιη, έξυπνη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Και το επιχείρημα ότι κοστίζει πολύ σημαίνει ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη καθόλου τι δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορεί να βάζει κανείς τιμές στα ανθρώπινα δικαιώματα ή στην ανθρώπινη ύπαρξη, ακόμη και σε πλούσιες χώρες όπως η Σουηδία. Ακούμε ότι είναι πολύ ακριβό το να συμπεριληφθούν τα άτομα με αναπηρίες. Εγώ πιστεύω ότι στο δικό μας κίνημα στη Σουηδία για τα άτομα με αναπηρίες ε, επικοινωνήσαμε με τον Νταν Άντρεσον, οικονομολόγο, ο οποίος κοίταξε, εξέτασε τα κέρδη που θα μπορούσε να αποκομίσει η κοινωνία. Όπως έγινε και σε άλλες μελέτες, σε άλλες χώρες, ο Νταν Άντερσον καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η προσβασιμότητα αποφέρει ωφέλη και οικονομικά. Είναι εποφελές το να συμπεριληφθούν όσο γίνεται περισσότεροι και το κόστος συμπερίληψης των ανθρώπων είναι πολύ χαμηλότερο από το κόστος αποκλεισμού τους. Αν κοιτάξει κανείς ε, το εισόδημα που δίνεται σε άτομα που συμμετέχουν στον κόσμο της εργασίας. Εγώ θα έλεγα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι χρειάζεται να αξιοποιήσουμε πλήρως αυτά τα συμπεράσματα. Πρέπει να τα εφαρμόσουμε στην πρακτική. Ζούμε σε εποχές κρίσης αυτής της στιγμής. Και αυτή είναι η κατάλληλη εποχή να επενδύσουμε για το μέλλον. Σε εποχές ε, ύφεσης, ε, χαμηλών ρυθμών ανάπτυξης, θα πρέπει να δείξουμε θάρρος, να πολεμήσουμε για τα ίσα δικαιώματα, την ίση αξία του καθενός και θα πρέπει να επιταχύνουμε τι προσπάθειές μας για να έχουμε μέτρα τα οποία θα προωθήσουν την προσβασιμότητα. Δεν μπορεί να βάζει κανείς ε, τιμή να τιμολογεί τα δικαιώματα των ανθρώπων να συμμετέχουν στην κοινωνία. Θα χρειαστεί λοιπόν να αντιληφθούμε, να ευαισθητοποιηθούμε στο γεγονός ότι αυτό θα αποφέρει ωφέλη για όλους. Εμείς ε, θα συμβάλλουμε γραπτά που τα οποία θα, και το κείμενο αυτό θα θέλαμε να επισυναυθεί στα πρακτικά. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα παρακαλέσω κάθε μία και κάθε ένα από εσά να ε, τηρήσουν με ε, πειθαρχία το χρόνο ομιλίας που τους χορηγείται βλέπετε από τις οθόνες πως γνωσασμένοι. Και τώρα θα ακούσουμε από την Ιταλία τον εκπρόσωπο του Ιταλικού Φόρουμ των Αναπηριών, τον Μάσο Ντανίελε, και παρακαλώ τον εκπρόσωπο της Αυστρίας, από το Αυστριακό Συμβούλιο Αναπηριών, την κυρία Μπέρναντετ Φερστάιντ να λάβει, να ετοιμάζεται να λάβει το λόγο επόμενη. Σε αυτή τη φάση της συζήτησης ε, καθίσταται αρκετά δύσκολο να πει κανείς κάτι πρωτότυπο. Παρ' όλα αυτά είμαστε εδώ για να καταγγείλουμε στεναρά την απόλυτη εγκατάλειψη των κοινωνικών πολιτικών υπέρ των ατόμων με αναπηρίες εκ μέρους της Ιταλικής κυβέρνησης. Η αρχή του τίποτα για εμάς χωρίς εμάς ε, έχει ανατραπεί. Όλα τα ρίχνουν πάνω μας χωρίς εμείς να συμμετέχουμε. Χωρίς εμάς η κυβέρνησή μας ε, έχει υποβαθμίσει το κοινωνικό κράτος, μείωσε τα κονδύλια για τις κοινωνικές πολιτικές, ε, για την αυτονομία, για την απασχόληση των ατομών με αναπηρία, για την εθελοντική ε, πολιτική υπηρεσία χωρίς εμάς υποβάθμισε τις διατάξεις για τους αναπήρους ε, τις φοροαπαλλαγές. Χωρίς εμάς ξεκίνησε μια άγρια εκστρατεία κατά των ε, αναπήρων ψευδών ή όχι, οι οποίοι θεωρήθηκαν υπεύθυνοι ότι εμπόδισαν την ανάπτυξη της χώρας μας. Και όλα αυτά αφού υπέγραψε και επικύρωσε τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών και αφού δημιούργησε έναν οργανισμό για την υλοποίησή της και την παρακολούθησή της. Δεδομένων όλων αυτών, εμείς κάνουμε έκκληση προς το Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να υπερασπίσουν τα δικαιώματα των αντόμων με αναπηρίες. Επ' αυτού η παρέμβαση του Προέδρου του Κοινοβουλίου μας καθησύχασε μάλλον σήμερα το πρωί. Το να θεωρούμε ότι ευθύνονται τα άτομα με αναπηρία για την οικονομική κρίση είναι κάτι άδικο, ανήθικο και παράνομο. Εμείς θέλουμε να αντιστραφεί η τάση κατά 360 μοίρες. Θέλουμε να γίνουν επενδύσεις στα άτομα με τις ε, με αναπηρίες ε, γιατί αν αυτοί ευημερούν θα ευημερήσει όλη η Ευρώπη θα, τα εισοδήματα των αναπηρών θα βοηθήσουν στην οικονομία της Ευρώπης ολόκληρου του πλανήτη για να επιτευχθεί αυτή η κοινωνική επανάσταση. Δεν χρειάζεται να επανεφεύρουμε τον τροχό. Αρκεί να ανακαλύψουμε την έννοια της αλληλεγγύης και να τη χρησιμοποιήσουμε για να υπερασπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αλληλεγγύη αποτελεί ακρογωνία ολίθο της μεσογειακής, του μεσογειακού πολιτισμού. Εμείς ελπίζουμε ότι από σήμερα στο εξή ο άνθρωπος, ο αξιοπρεπής άνθρωπος θα αποτελέσει τον ακρογωνίων, ολίθο οποιασδήποτε κοινωνική πολιτική. Και είμαστε εδώ για να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση και να τρέφουμε αυτή την ελπίδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο συνάδελφος από την Αυστρία. Bernadette Φορεστάιν. Επίσης, οι ευρωβουλευτές Νίλς Τόρβανσον πρώτα απ' όλα να προετοιμαστεί για να πάρει το λόγο μετά. Παρακαλώ η Αυστρία τώρα. Jelezték, Από ό,τι φαίνεται δεν είναι εδώ ο συνάδελφος. Νίλ Στόρβανσον τότε. Και μετά Σοπάλ να ετοιμάζεται την επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και καλησπέρα σας. Στην καθημερινή μου ζωή έξω από το Κοινοβούλιο είμαι επικεφαλής της οργάνωσης για, τους, για τα άτομα με αναπηρία πνευματική και σωματική και λέω διανοητική αναπηρία και λέμε ότι έχουμε το μήνυμα, το κύριο μήνυμα να μεταδώσουμε ότι κανείς δεν έχει επιλέξει να έχει τέτοια αναπηρία. Όταν με ρωτάει κανείς τι κάνει ο γιος σου, ε, πάντα τους απαντάω ποιον από όλους. Λες, εγώ έχω τέσσερα παιδιά. Βέβαια εννοούν τον ε, πρώτο μου γιο, τον Λίνους. Όμως εγώ εδώ έχω έρθει για να σας μιλήσω για τον Κρίστοφερ, τον τρίτο γιο μου. Ο Κρίστοφερ είναι παιδί του συνδρόμου Κλίνεφελτ Αντί δηλαδή να έχει χρωμόσωμα X, Χ, Y, έχει χρωμόσωμα Χ, Χ, Y, διπλό X και Y. Αυτό σημαίνει ότι έχει διανοητικά προβλήματα και άρα η δυνατότητά του για να βρει, δυνατότητες του να βρει θέση εργασίας είναι ισχνές και πολύ πιο ισχνές, γίνονται όλο και πιο ισχνές όσο αυξάνεται το ποσοστό ανεργίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε να κάνουμε ποσοστά ανεργία στις περισσότερες από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης καταστροφικά και ιδιαίτερα κακά στις χώρες με κρίση που καθιστούν αδύνατη τη διαφύλαξη της ε, ευημερία και του, καθε... του κοινωνικού κράτους πρόνοιας όπως το γνωρίζαμε εμείς τουλάχιστον στη Φιλανδία. Έτσι λοιπόν θα υποφέρουν τα άτομα με αναπηρία περισσότερο από το κάθε ένα και γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε, διότι οι συνέπειες του να χάσουμε αυτόν τον αγώνα κατά της ε, απομόνωσης του αποκλεισμού είναι φρικτές. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα παρακαλώ να λάβει το λόγο ο κύριος Σουτ Πάλ από την Ουγγαρία και να ετοιμάζεται η Μαριάν Χάρκιν, συνάδελφος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα είναι η επόμενη. Παρακαλώ τώρα λοιπόν. Πάλ Σουτ. Ευχαριστώ. Η κρίση και η επίλυση της κρίσης είναι κάτι για το οποίο μιλάει ο κόσμος. Συνήθως μιλάει για την εκπαίδευση, την απασχόληση. Το πραγματικό μου ζήτημα είναι έχουμε πλήρη πρόσβαση στα αγαθά αυτά ή υπάρχουν τελικά εμπόδια στο δρόμο μας όταν πρόκειται για την εκμάθηση ή για την εργασία. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα πραγματικό ευρωπαϊκό πλαίσιο ώστε να έρθουν τα εμπόδια αυτά, να τα υπερπηδήσουμε, να τα ξεπεράσουμε. Πρέπει να είμαστε σαφείς για το τι μπορεί να κάνει ο κόσμος και τι δεν μπορεί. Όσον αφορά και την απασχόληση, πρέπει να υποστηρίξουμε όλες τις οικονομικές και τις κοινωνικές λύσεις, οι οποίες έχουν ξεκινήσει, αλλά πρέπει να αναπτυχθούν παρετέρω. Πρέπει να φτιάξουμε δίκτυα, διότι δεν χρειαζόμαστε ανταγωνισμό σε αυτή την περίοδο κρίσης, όχι. Πρέπει να βάλουμε τις δυνάμεις μας μαζί. Πέρα από την άρση των εμποδίων πρέπει χέρι-χέρι να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη τεχνολογίας που μας βοηθάει. Οι περισσότεροι από εμά τη χρειαζόμαστε αυτή την ανάπτυξη της τεχνολογίας, γιατί μόνο έτσι με την τεχνολογία μπορούμε να συμμετέχουμε πλήρως στην καθημερινή ζωή στην κοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστώ που λάβατε υπόψη σας και το χρόνο. Τώρα η Μαριάν Χάρκιν έχει το λόγο. Και πριν να αρχίσετε, να σας πω η Λία Σέφερτ από τη Γερμανία να ετοιμάζεται να πάρει το λόγο αμέσω μετά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σήμερα το απόγευμα συζητούμε για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών, σήμερα που είμαστε σε περίοδο κρίσης. Τώρα για όλους τους πολίτες, αλλά κυρίως εκείνους με αναπηρίες, αυτοί που βρίσκονται δηλαδή στο περιθώριο για κάποιο λόγο, η κρίση και ιδιαίτερα μια οικονομική κρίση μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Τα ακούσαμε και από τους συναδέρφους από την Ιταλία, από την Τσεχία, από την Ελλάδα. Ακούσαμε τις επιπτώσεις αυτές και πρόκειται για χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπετε ότι η κρίση έχει ανατρέψει την κοινωνική πρόοδο, την έχει πάει πίσω, γιατί τώρα επικεντρωνόμαστε στην οικονομική κατάσταση μόνο βλέπουμε πόσο αρνητικές επιπτώσεις έχει στην ποιότητα ζωής, γιατί γίνονται περικοπές στις υπηρεσίες. Τι θα κάνουν όμως οι οικογένειες, ε, τα άτομα που υποφέρουν. Με περιορισμένους πόρους η ζωή τους γίνεται πολύ δύσκολη. Δεν έχουν ε, κοινωνική βοήθεια, δεν έχουν κοινωνικές υπηρεσίες και για ανθρώπους με αναπηρίες καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για μια πραγματικά προσωπική τραγωδία, γιατί δεν μπορούν πια να ζουν ανεξάρτητα, πρέπει να εξαρτώνται από τους άλλους, δεν είναι πια αυτόνομοι. τι νόημα έχει να μιλάμε για την ελευθερία διακίνησης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν τα άτομα δεν μπορούν να έχουν κάποια βοήθεια. Την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε την ετήσια μελέτη που έδειξε μια πολύ συχνή εικόνα για την Ευρώπη. Και υπάρχει κάτι που ονομάζουμε Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το οποίο δείχνει την πρόοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την κατεύθυνση των στόχων του 2020. Δυστυχώς όμως η έκθεση αυτή η πρόοδου βρίσκεται αντιμέτωπη, μάλλον ε, περιλαμβάνει οικονομικούς δείκτες, μιλάει για προγράμματα σταθερότητας και ανάπτυξης, αλλά δεν υπάρχουν δείκτες για τα κοινωνικά αγαθά, ούτε για τις ε, κοινωνικές επιτυχίες ή τη λιτότητα από την άλλη μεριά. Συνεπώς, τα μειονεκτήματα μένουν αόρατα. Εμείς από την κρίση αυτή πρέπει να προχωρήσουμε με διαφορετικό τρόπο, να βγούμε δηλαδή με άλλη νοτροπία από αυτήν με την οποία μπήκαμε. Αν συνδέσουμε τις οικονομικές πολιτικές και τις, ε, τα κοινωνικά αποτελέσματα και τα λάβουμε υπόψη μας τις οικονομικές μας επιπτώσεις, αυτό θα κάνει ήδη μια μεγάλη διαφορά. Ευχαριστούμε. Τώρα το λόγο έχει ο Ηλία Σάιφερ από τη Γερμανία και να ετοιμάζεται ο εκπρόσωπος της Ιταλίας από το Ιταλικό ε, Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρίες. Σήμερα πολλά υπόθηκαν, πολλά σωστά και εύστοχα σχόλια υπόθηκαν. Δεν θέλω να επαναλάβω, θα προσθέσω μόνο δύο πράγματα. Πρώτον, σήμερα Συζητούμε διαρκώ λέγοντα ότι βρισκόμαστε σε άμυνα, ότι αμυνόμαστε σε έναν αγώνα με ανθρωπιστική κρίση. Πρέπει ωστόσο να επισημάνουμε ότι η Σύμβαση των Ανθρωπινών Δικαιωμάτων των, ε, δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία των Ηνωμένων Εθνών είναι μια σύμβαση επέκταση των δικαιωμάτων και προστασία των ε, ατόμων ε, με ή χωρί αναπηρία. Δεύτερον, πρέπει να πούμε ότι η Ευρώπη ξεπερνάει τα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, αν θέλουμε να προχωρήσουμε, δεν είναι δυνατόν να επιτρέπουμε τα κράτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως οι παραδείγματι τα κράτη που ανήκαν στο παρελθόν στην ε, Σοβιετική Ένωση, τα κράτη της Βαλκανικής, να παραμένουν στο περιθώριο και πάνω απ' όλα να μην έχουν ε, αρκετή πρόοδο στον τομέα αυτών. Ε, τρίτον, η Γερμανία συχνά επικρίνεται για το γεγονός ότι δεν έχει ε, επιτρέψει την πρόοδο της πέμπτης διακρί... Ε, οδηγίας κατά των διακρίσεων η γερμανική κυβέρνηση. Αυτό είναι αλήθεια και ντρεπόμαστε όλοι γι' αυτό, αισθανόμαστε ε, όνειδος, αλλά πρέπει να πω ότι όλα τα άτομα με αναπηρία και όλες οι οργανώσεις μας στη Γερμανία αγωνίζονται για την προαγωγή αυτής της οδηγίας, της πέμπτης οδηγίας για τις διακρίσεις κατά των διακρίσεων και θα πιέσουμε την κυβέρνησή μας να την προωθήσει. Επίσης θέλω να επισημάνω ότι ε, επειδή μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί και επειδή αποδεχόμαστε ότι είμαστε διαφορετικοί, μπορούμε να συνεργαζόμαστε μεταξύ μας. Αυτό είναι μια αρχή η οποία πρέπει να υλοποιηθεί σε ολόκληρη την κοινωνία, όχι μόνο μέσα στο κίνημα των ατόμων με αναπηρία. Εάν τα καταφέρουμε αυτά, τότε θα έχουμε καταφέρει πάρα πολύ σημαντική πρόοδο για όλε τι κοινωνίε μα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ για τα σχόλιά σας. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τον Ιταλό συνάδελφο Τριτσιόνε να λάβει τον λόγο. και να ετοιμαστεί η Γαλλίδα εκπρόσωπος με την ποιότητα για να λάβει τον λόγο μετά. Ευχαριστώ τους ευρωβουλευτές που είναι παρόντες. Τα άτομα με αναπηρίες αποτελούν πόρο, όχι δαπάνη. Πρέπει να εκφραστούμε όσο μπορούμε καλύτερα και να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Το να μην μπορούμε να ζούμε έτσι αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και απώλεια για ολόκληρη την ανθρωπότητα, η οποία δεν μπορεί να υποφεληθεί από τη δική μας συμβουλή, αλλά και απώλεια οικονομική. Και αυτό μπορεί να υπολογιστεί με νούμερα. Εμεί είμαστε η ευκαιρία για να βγούμε από την οικονομική κρίση. Πρέπει να επενδύσετε σε εμά. Οι περικοπέ ε, κονδυλίων όχι μόνο παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη συνθήκη, αλλά χάνουμε περισσότερα χρήματα από όσα θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε. Το να στηρίσουμε ένα παιδί με αναπηρίε από την κατάλληλη παιδεία, το μεταμορφώνουμε σε έναν ενήλικο εξαρτημένο. Τεράστιο κόστος λοιπόν για την κοινωνία η οποία θα πρέπει να καταβάλει χρήματα σε προσωπικό που θα το παρακολουθεί καθημερινά. Επιπλέον οι συγγενείς, ειδικότερα οι μητέρες, πρέπει να εργάζονται λιγότερο ώστε να προσέχουν να φροντίζουν την ε, οικογένειά τους, τα μέλη της οικογένειάς τους με αναπηρία. Μιλάμε για άτομα που βγαίνουν από την αγορά εργασίας. Άλλο ένα λοιπόν κοινωνικό κόστος. Τα άτομα με αναπηρίες είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού που δεν συμμετέχει ακόμα στην αγορά εργασίας. Με την κατάλληλη παιδεία, με κατάλληλες παρεμβάσεις μπορούν να επιτύχουν αυτονομία, ανεξαρτησία για την υπόλοιπη του ζωή συμμετέχοντας στο χώρο εργασίας, αποτελώντας ε, όφελος για την κοινωνία. Ένα σχόλιο για την πρώτη ολομέλεια, το άρθρο 12 της συνθήκης αφορά την ίση αναγνώριση της νομικής ικανότητας ενώπιον του νομού. Τι συμβαίνει όταν ένα άτομο με αναπηρία δεν μπορεί να ασκήσει τα δικά του νομικά δικαιώματα γιατί δεν μπορεί να μιλήσει, να κατανοήσει ή να επικοινωνήσει στο επίπεδο που απαιτείται για να συζητήσει ζητήματα νομικά. Η συνθήκη ορίζει ότι όσοι χρειάζονται υποστήριξη θα πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους ένα σύστημα υποστήριξης Όπω συμβαίνει και για τον αυτισμό, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναγνωρίσει ότι όλε οι μορφέ επικοινωνία που έχουν επικαιρωθεί επιστημονικά μπορούν να ισχύουν για την επικοινωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Από τη Γαλλία τώρα η Μαρή Διπιότ. Και θα ήθελα να στήσω από την Ισπανίδα συναδέλφο Άρμα Ιωάννης ε, Λουίς Μανιάτ να ετοιμαστεί να μιλήσει στη συνέχεια. Καλημέρα. Είμαι πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών για Δράση που αγωνιζόμαστε κατά οποιασδήποτε διάκρισης, ειδικότερα κατά της διπλής διάκρισης που βιώνουν οι γυναίκες με αναπηρία. Θα σας μιλήσω σήμερα για τις γυναίκες. Θέλουμε, θέλω να λάβουμε υπόψη τις περιπτώσεις βίας που υφίστανται γυναίκες με αναπηρία 36% των γυναικών στη Γαλλία, 72% των γυναικών με αναπηρία πέφτουν θύματα και θέλω αυτές οι διακρίσεις να σταματήσουν κατά των γυναικών με αναπηρίες και να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Αυτές οι περιπτώσεις βίας είναι σωματικές όσο και ηθική παρενόχληση και βιασμός. Οι γυναίκες με αναπηρία ε, είναι κλεισμένοι σπίτια τους και δεν μπορούν να διαμαρτυρηθούν, δεν μπορούν να το καταγγείλουν. Το δεύτερο που θέλω να καταγγείλω είναι η υγεία. Οι γυναίκες με αναπηρία, τουλάχιστον στη Γαλλία και πιστεύω και σε πολλές άλλες χώρες, δεν λαμβάνουν τις απαραίτητες φροντίδες. Σημαίνει ότι ελάχιστες ε, γυναικολογικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες και το να είναι μια γυναίκα με αναπηρία μητέρα σήμερα θεωρείται σαν να είναι κάποιος άνθρωπος που κάνει λάθος. Οι γυναίκες με αναπηρία κάθε μέρα πρέπει να αγωνίζονται για να γίνουν σεβαστές ως πολίτες. Αυτό που θα ήθελα να καταγγείλω επίσης είναι ότι αν θέλουμε η κρίση να περάσει, αν θέλουμε να βγούμε από την κρίση, πρέπει οι γυναίκες να είναι παρούσες παντού. Ότι οι γυναίκες με αναπηρία θα πρέπει να έχουν τη θέση τους σε όλες τις επιτροπές. Οι γυναίκες με αναπηρία θα πρέπει να ακουστούν να συμμετέχουν στην κοινωνία. Είμαστε πολίτες εξ ολοκλήρου. Έχουμε δικαιώματα, έχουμε ανάγκες και μαζί οι γυναίκες και οι άντρες θα αλλάξουμε το βλέμμα προς τις διαφορές. 22% των αναπήρων γυναικών στη γυναίκα μόνο βρίσκουν ε, ε, εργασία σε σύγκριση με 46% των αντρών. Και εκεί έχουμε λοιπόν διακρίσεις σε θέματα φύλου. Ζητώ λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε όλες τις επιτροπές να μεριμνήσουν ώστε οι γυναίκες με αναπηρία να είναι παρούσες σε όλες τις συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα Ισπανία. Γιάννης Λουίς Μονβάλ. Και μετά ο επόμενος ομιλητής, ο Πίτερ Λάμπρεχτ, να ετοιμάζεται. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρου ε, του Συμβουλίου Εκπροσώπων Ατόμων ε, με Αναπηρίες ω Αντιπρόεδρο τη Ισπανική Ομοσπονδία Ασπανίων Ασθενειών, θέλω να σα ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να έρθω και να σα μιλήσω. Όπως ακούσαμε ήδη, πρέπει και να το επαναλαμβάνουμε, η οικονομική κρίση επηρεάζει πάρα πολύ σοβαρά αυτούς που περισσότερο έχουν ανάγκες, δηλαδή τα άτομα με αναπηρίες, τους επαγγελματίε που ασχολούνται μαζί του και τις οικογένειε τους. Και είναι μέγα σφάλμα να πληρώνουν την κρίση εκείνοι που φταίνουν λιγότερο για αυτή. Εκείνοι που περισσότερο έχουν ανάγκες χάνουν μέρος των εσόδων τους, μέρος της φροντίδας που δικαιούνται. Στην πραγματικότητα όμως πλήττονται τα ίδια τα θεμέλια της κοινωνίας. Όπως ακούσαμε και πριν, η αναπηρία δεν σημαίνει μόνο ε, αναπηρία φυσική ή διανοητική, σημαίνει και μοναξιά. Και αυτό είναι που είναι κρίμα, η μοναξιά. Η ελευθερία και η αξιοπρέπεια στην κοινωνία μας πρέπει να διασφαλίζεται από τους δημοκρατικά εκλεγμένους ηγέτες. Όμως οποιαδήποτε κυβέρνηση που θέλει να διασφαλίσει την ελευθερία και την αξιοπρέπεια πρέπει να είναι ίδια ελεύθερη και αξιοπρεπής. Με τη στήριξη του λαού έχει εκλεγεί εξάλλου αλλά τελικά μάλλον δίνουν την προτεραιότητα στις αγορές και στην οικονομία οι οποίες ε, λειτουργούν ανασταλτικά και τελικά ε, πιέζουν πάρα πολύ τους πιο αδύναμους και τους βάζουν σε ακόμα, χειρότερη θέση. Έτσι λοιπόν πρέπει να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει. Το θέμα δεν είναι να λέμε λόγια, είναι και να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ειδών κακά. Το ένα είναι οι χρόνιες ασθένειες και αναπηρίες. Έχασα πριν από έξι μήνες το γιο μου 8 ετών. Το άλλο όμως είναι πώς θα το αποφύγουμε. Και θα το αποφύγουμε αν ο καθένας παίξει το ρόλο του. Οπότε σας ευχαριστώ όλους εσάς που παίζετε το ρόλο σας σε αυτή την υπόθεση αλλά όχι εκείνους οι οποίοι το λένε αλλά δεν το κάνουν. Οι κάλπες είναι αυτές όμως που θα δείξουν ποιος τελικά πραγματικά ε, φέρει σε πέρα στο ρόλο του και ποιος όχι. Ευχαριστούμε. Τέλος. Πίτερ Λάμπρεχτ. Ονομάζομαι Πίτερ Λάμπρετς από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ανεξάρτητης ε, Διαβίωσης. Ως οργάνωση βάσης με μέλη σε όλη την Ευρώπη καταγράφουμε την πολύ ανησυχητική εξέλιξη από την κρίση εξ αρχής. Ε, κρούμε τον ε, κόδωνα του κινδύνου απευθυνόμενοι σε βουλευτές, ευρωβουλευτές, ανεξάρτητες οργανώσεις ευρωπαϊκές και ε, επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε για την κοινωνία των πολιτών τη δραστηριοποίηση που χρειάζεται τόσο στην Ευρώπη αλλά και στη διεθνή σκηνή όπως κάνουν και οι διεθνείς μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Πρέπει το θέμα αυτό να μπει στην ημερήσια διάταξη, να προαχθεί καθώς έχει αποδειχθεί και με πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα ότι είναι ήδη καταστροφικές οι συνέπειες, καταστροφικές οι συνέπειες της κρίσης. Από το να κρούμε λοιπόν τον κόδωνα του κινδύνου υπάρχει τίποτα άλλο να κάνουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευαισθητοποιήσουμε του αρμόδιους για τη χάραξη τη πολιτική, αλλά και την κοινή γνώμη. Αυτό κάνουμε ιδιαιτέρω. Η δική μα οργάνωση, το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Αναπηριών και πολλέ άλλε. Ε, οργανώσεις, όμως μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα ακόμη. Η δική μας η οργάνωση για την ανεξάρτητη διαβίωση έχει, επί παραδείγματι, βοηθήσει στη σύνταξη του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν είναι το ίδιο κείμενο που ονομάζεται το ψήφισμα και που συζητιέται σήμερα. Ε, είναι στόχος μας να προωθήσουμε όμως ένα ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σε αυτό επιδιώκουμε τη συνεργασία με ευρωβουλευτές για να ε, συνομιλήσουμε μαζί τους, να ακούσουμε και να δεχθούμε συμβουλές, να δώσουμε συμβουλές και ταυτόχρονα να προωθήσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συνομιλούμε με μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προκειμένου να προβλεφθεί το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη τη ε, συνεδρίασης τη Επιτροπή, με μια προφορική ερώτηση από τι εργασίε τη Επιτροπή Απασχόληση και να εξασφαλιστεί έτσι πρόοδο ε, του ζητήματο μέχρι τελική υιοθέτηση από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του σχετικού ψηφίσματο. Είναι στόχο ε, ίσω πολύ απαιτητικό για μια οργάνωση μικρή όπω η δική μα, όμω εργαζόμαστε σκληρά, συνεργαζόμαστε και έχουμε τη στήριξη και άλλων κυβερνητικών οργανώσεων αλλά και πολιτών. Και θα ήθελα επί τη ευκαιρία αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Ατόμων με Αναπηρία να σα ενημερώσω για τι προσπάθειέ μα. Μπορώ να σα δώσω επίση, εάν θέλετε, επιπλέον πληροφορίε που μπορούν να προσαρτηθούν στην έκθεση των σημερινών εργασιών, ε, γιατί ζητούμε την υποστήριξη των πάντων όλοι εσάς όσοι εκπροσωπείτε οργανώσεις ατόμων με αναπηρία θα θέλαμε να ζητήσετε από τον βουλευτή σας, από τον ευρωβουλευτή σας, από τον εκπρόσωπο στην περιοχή σας ή την πόλη σας να υποστηρίξει την πρωτοβουλία αυτή. Σας ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που μας δίνετε. Θέλουμε δικαιώματα και όχι ελεημοσύνη. Ευχαριστώ. Köszönöm, gondolom, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι μπορούσαμε να κλείσουμε με ομιλία πιο εύστοχη και πιο εύγλωτη από αυτή που μόλις ακούσαμε. Χρειαζόμαστε μέτρα, χρειαζόμαστε πρωτοβουλίες. όπου οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία και τις οργανώσεις τους κάνουν δουλειά μαζί, γιατί μόνο αν δουλεύουμε μαζί μπορούμε να επιτύχουμε. Τώρα φτάνουμε στο δεύτερο τμήμα, λοιπόν. Ε, ολοκληρώνουμε το δεύτερο τμήμα τη απογευματινή συνεδρία σα. Σα ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κατά λίγο ξεπεράσει το χρόνο μα, αλλά πάντω όχι πολύ. Όχι πολύ και τώρα νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε για το τρίτο κύκλο παρουσιάσεων. Πρώτο όμω θα κάνουμε μια προβολή ταινία. Και συγκεκριμένα βίντεο ε, μαγνητοσκοπημένου μηνύματος του κύριου Φαν Ρόμποη, Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ας τον ακούσουμε. Ε. Γιατί σου κάτσε κάνεις με βλακική. Τι μας έχουν γαμίσει μην. Τι θες να Κλείστε μικρό. Elnézést kérünk a technikai probléma miatt. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα από ό,τι φαίνεται που προσπαθούμε να λύσουμε. Λίγο υπομονή παρακαλώ. Λοιπόν, περιμένουμε να λυθεί το τεχνικό πρόβλημα. Προσπαθούμε. Πάντως, οι συμμετέχοντες στο τρίτο πάνελ, αυτοί που θα προεδρεύσουν, να έρθουν παρακαλώ να πάρουν τις θέσεις τους εδώ, στο Προεδρείο. Buenas tardes A todos y a todas. Καλησπέρα. Βρισκόμαστε στην, στο τρίτο τμήμα των εργασιών του Ευρωπαϊκού Αυτού Κοινοβουλίου Ατόμων με Αναπηρίες. Είμαι η Άννα Παλαέθ από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Φόρου Ατόμων με Αναπηρίες και εκπροσωπώ επίσης και την Επιτροπή Γυναικών. Είμαι συμπρόεδρος σε αυτό το τμήμα της συνεδρίασης με έναν από τους ε, αντιπροέδρους της διακομματικής ε, ομάδας, ο κ. Γκοβάντι που θα έρθει σε λίγο. Μου λένε, λέει η κυρία Πελάιφ, ότι μας έχει μείνει από σήμερα το πρωί το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα του Πρόεδρου του Συμβουλίου, του κ. Φανρομπάη. Θα τον ακούσουμε τώρα, ευθύς αμέσω λοιπόν. Και μετά θα σας δώσουμε το λόγο πρώτα απ' όλα στον κ. Βαρδακαστάνη, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρίες, για να αντιδράσει στο μήνυμα αυτό. Λοιπόν, ας ακούσουμε τον κύριο Φανρομπάη. persons with disabilities. Our... Οι δράσεις μας για την αποκατάσταση της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης ε, επικεντρώνονται στο να διατηρήσουμε ζωντανό το κοινωνικό μας μοντέλο, ένα μοντέλο με στόχο την ευημερία 500 εκατομμυρίων ανθρώπων, διότι η Ευρώπη είναι ένα έργο αξίας και ανθρώπων, ένα έργο με καρδιά. Σας εύχομαι επικοδομητικές συζητήσεις σήμερα. <laughs> Νομίζω ότι ακούσαμε μόλις το τελευταίο τμήμα. Μήπως γίνεται να το ακούσουμε από την αρχή το μήνυμα σας παρακαλώ. Νομίζω ότι πάλι έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με το βίντεο. Μέχρι να λυθεί. Ας αρχίσουμε. Το τμήμα αυτό είναι αφιερωμένο στην ελεύθερη κυκλοφορία και την ιδιότητα του πολίτη των ατόμων με αναπηρίες. Υπάρχουν ακόμα εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν και αυτό θέλουμε να δούμε. Πώς θα ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια που μας δυσκολεύουν να χαρούμε πλήρως τις ιδιότητάς μας ως πολίτες και τις ελευθερίες διακίνησης. Σήμερα το πρωί η Σέρμη από την ε, Ισπανία ήρθε. Το πρωί, πρωί-πρωί από την Ισπανία. Λοιπόν, όταν φτάσαμε, μάθαμε ότι ένας από τους ε, συναδέρφους που ερχόταν ε, σαν εμπειρική καρέκλα, η υπηρεσία, η αρμόδια για την μειωμένη κινητικότητα, είχε ξεχάσει στο αεροδρόμιο την ε, αναπηρική του καρέκλα. Οπότε έφτασε εδώ στις Βρυξέλλες χωρίς να έχει το βασικό του, αυτό που του ήταν αναγκαίο για να μπορεί να μετακινηθεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν, θα συμφωνήσετε μαζί μου πόσο σοβαρό είναι αυτό. Και γιατί πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προκειμένου να μπορούν να επωφεληθούν από την ελευθερία διακίνησης. Και αυτά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Μια περιοχή του κόσμου η οποία κύρωσε μόλις για πρώτη φορά μια σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Σε ένα γεωγραφικό χώρο όπου 24 από τις 26 χώρες μέλη έχουν ήδη κυρώσει τη σύμβαση αυτή. Μια σύμβαση η οποία ζητάει μέτρα, υπευθυνότητα από πλευράς των χωρών μελών, από τους ηγέτες, από τις κυβερνήσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν ακριβώς αυτά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ανθρώπινα δικαιώματα και των ατόμων με αναπηρίες. Στη σύμβαση αυτή η προσβασιμότητα αποτελεί μία από τις βασικές αρχές για να διασφαλιστούν ακριβώς αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρόκειται για ένα μέσο το οποίο θα πρέπει οριζόντια να ισχύει σε όλες τις πολιτικές και σε όλα τα μέτρα που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες μέλη. Και εκείνες δηλαδή που έχουν ε, κυρώσει τη σύμβαση. Η προσβασιμότητα αποτελεί την αρχή η οποία θα εξασφαλίσει την εφαρμογή των δικαιωμάτων αυτών των ατόμων με αναπηρίες. Έτσι λοιπόν η σύμβαση στο άρθρο 9 λέει ποιος είναι ο κύριος στόχος της προσβασιμότητας είναι τα άτομα με αναπηρίες να μπορούμε να ζούμε αυτόνομα. Όπου, με όποιον και όπως θέλουμε. Να μπορούμε να συμμετέχουμε επίσης πλήρως σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας. Στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην υγεία, στη, στον πολιτισμό, στην ψυχαγωγία και στην πολιτική ζωή βέβαια. Η σύμβαση είναι απόλυτα σαφής για το τι πρέπει να κάνουν τα κράτη-μέλη που την έχω δηλαδή συνυπογράψει για να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους. Λέει πολύ συγκεκριμένα να λαμβάνουν όλα τα μέτρα που χρειάζεται για να διασφαλίζουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες υπό ίσες όρες στην πληροφορική, στον ε, περίγυρο, στην επικοινωνία, στα αγαθά, στις υπηρεσίες, παντού, σε όλα αυτά. Όμως, τηρείται η σύμβαση αυτή. Ισχύει. Είμαστε, ζούμε όντως επίσης ώρες με τους άλλους. Χαίρομαι των ε, θεμελιών αυτών ελευθεριών. Φαντάζομαι ότι και εσείς συμφωνείτε μαζί μου ότι η απάντηση είναι πολύ σχετική. Τα άτομα με αναπηρίες προς το παρόν δεν μπορούμε να υποφεληθούμε πλήρως από τα πραγματικά μας δικαιώματα. Το δικαίωμα στην ελεύθερη κυκλοφορία διαπιστώνουμε ότι έχουμε εμπόδια σε όλους τους τομείς της ζωής. Και οι συνθήκες προσβασιμότητας είναι πολύ διαφορετικές. Όχι μόνο από χώρα σε χώρα, αλλά και μέσα στην ίδια χώρα υπάρχουν τεράστιες διαφορές και μέσα στην ίδια περιφέρεια. Εμείς θέλουμε ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων με αναπηρίες. Μεταφορές, για παράδειγμα, σας τα είπε και ο συνάδελφος σήμερα το πρωί δυσκολευόμαστε να χρησιμοποιήσουμε κάποια προϊόντα. Κινητά τηλέφωνα, για παράδειγμα. Επίσης, βρισκόμαστε μπροστά σε εμπόδια όταν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες. Έχουμε εξίσου πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, τις κοινωτικές υπηρεσίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης όρες ή στις χώρες μας στις πόλεις μας. Οπότε, αν θυμόσαστε τη δημοσίευση που κάναμε πέρυσι από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα άτομα με αναπηρίες που μιλούσε για την ελευθερία κυκλοφορίας και διακίνησης, θα θυμόσαστε τα κενά που εντοπίσαμε και που παραμένουν δυστυχώς όσον αφορά την πρόσβαση στα αγαθά και στις υπηρεσίες κάτι το οποίο μας εμποδίζει να χαρούμε και να επωφεληθούμε από τα δικαιώματά μας επίσης ώρες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν έχει τρεις πρωτοβουλίες, σημαντικές πρωτοβουλίες. Έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα. Είναι η Ευρωπαϊκή Πράξη για την Προσβασιμότητα που αναφέρθηκε σήμερα. Πόσο θα πρέπει να περιμένουμε ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πόσο θα μας κάνει ακόμα να περιμένουμε για να δεσμευτεί, που κανονικά έπρεπε να είναι για φέτος. Ελπίζουμε το Φεβρουάριο να το έχουμε. Το EDF είμαστε πεπισμένοι ότι χρειαζόμαστε αυτή την πράξη, μια φιλόδοξη πράξη, η οποία καλύπτει όλες τις πτυχές που αναφέρονται στη σύμβαση του ΟΗΕ στο άρθρο 9. Επίσης, αυτές τις μέρες Ξέρουμε ότι αυτό που εδώ και δύο χρόνια περιμένουμε, τη δημοσίευση της νομοθετικής πρότασης για την πρόσβαση στις δημόσιες ιστοσελίδες. Επιτέλους, υπάρχουν τόσες πληροφορίες, υπάρχουν τόσες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του διαδικτύου. Ε, λοιπόν, εμείς, τα άτομα με αναπηρίες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα δεν μπορούμε να αποφεληθούμε επίσης ώρες από τις υπηρεσίες αυτές που προσφέρονται μέσω διαδικτύου. Την Δευτέρα δημοσιεύθηκε η νομοθετική αυτή πρόταση και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ πιστεύει ότι θα χρησιμεύσει πραγματικά για να προωθηθούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Τέλος, θέλω να αναφέρω και την αναθεώρηση που γίνεται αυτή την εποχή όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Είναι στην εσωτερική αγορά που εξετάζεται αυτό το θέμα. Τι λέει λέει ότι είναι πολύ σημαντικός αυτός ο τομέας για την απασχόληση, για παράδειγμα, των ατόμων με αναπηρίες. Βλέπετε, του χρόνου είναι η Ευρωπαϊκή Χρονιά, το Ευρωπαϊκό Έτος για τους πολίτες. Πολίτες οι οποίοι κανονικά έχουν πάρα πολλά δικαιώματα. Τι γίνεται όμως με τα άτομα με αναπηρίες, έχουν τα ίδια. Πρέπει αν μη τι άλλο να αναγνωριστούν. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα, πάρα πολλοί πολίτες, γυναίκες και άντρες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν αναγνωρίζονται εξίσου από τον νόμο. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ως πολίτες είναι νεκροί. Δεν έχουν κοινωνικά πολιτικά δικαιώματα, δεν μπορούν να ψηφίσουν, δεν μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια, δεν μπορούν να ζήσουν όπου επιθυμούν, δεν μπορούν να έχουν τραπεζικό λογαριασμό, δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στη λήψη αποφάσεων. Πολλά λοιπόν μένουν ακόμα να γίνουν. Πάρα πολλά όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες, επίσης μεταξύ και γυναικών. Φανταστείτε τις γυναίκες με αναπηρίες. Φανταστείτε σε τι θέση βρίσκονται εκείνες. Το δικαίωμα να κάνουν παιδιά, το δικαίωμα στην υγεία, το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα και αυτόνομα. Ελπίζω σήμερα να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις, ιδέες που θα μας βοηθήσουν να χτίσουμε μια Ευρώπη πραγματικά χωρίς εμπόδια για τα άτομα με αναπηρίες. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Σύρπα Πετικάινεν. Μπερδεύομαι να προφέρω το όνομα, λέει ο Μιλήτρια. Σύρπα Πιέτη Κάινεν, που είναι αντιπρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Εσωτερική Αγορά και την ε, Προστασία του Πολίτη. Παρακαλώ, Σύρπα, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω για την προσβασιμότητα και πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το ζήτημα στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς εδώ στο Κοινοβούλιο. Πρώτα απ' όλα, πολύ σύντομα, θα ήθελα να αγγίξω δύο βασικές θεμελιώδεις ιδέες που συζητήθηκαν όλη την ημέρα σήμερα. Την έννοια των συνταγματικών δικαιωμάτων ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με συνταγματικά δικαιώματα τα οποία αντικειμενικά αποτελούν δικαιώματα. Εδώ τα βλέπουμε υπό συγκεκριμένο πρίσμα. Είναι κάτι το οποίο διασφαλίζεται, φυλάσσεται από τις συνθήκες. Είναι κάτι υποχρεωτικό. Είναι υποχρεωτικό για την Επιτροπή και για το Κοινοβούλιο στην νομοθεσία τους να λαμβάνουν υπόψη. Τα δικαιώματα αυτά δεν είναι εθελοντική πτυχή παρότι συχνά το ξεχνάμε. Δεύτερον, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τις προσπάθειές μας εδώ στο Κοινοβούλιο για την οδηγία κατά οποιασδήποτε μορφής διάκρισης. Πιστεύω ότι αυτός θα πρέπει να είναι ο απότερος στόχος, διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα οριζόντια ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία. και οποιονδήποτε ατόμων συνταγματικά και βασικά δικαιώματα. Η τρίτη γενική έννοια είναι η γενικότερη αρχή που αφορά ουσιαστικά οριζόντια όλους τους τομείς ε, και όλα τα ζητήματα για τα οποία συζητάμε εδώ είναι το ζήτημα των ε, περιβαλλόντων που παρέχουν δυνατότητες και της ανάληψης θετικών δράσεων μέσω της προσβασιμότητας. Δεν είναι μόνο λοιπόν το ζήτημα να αφαιρέσουμε τα εμπόδια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα είναι να πάμε ένα βήμα πιο μπροστά. Να δώσουμε τη δυνατότητα για θετικές δράσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ισότητα, στο να βρίσκονται τα άτομα με αναπηρία σε ίσο επίπεδο με όλους τους υπόλοιπους. Πού μας οδηγεί αυτό όσον αφορά δύο ζητήματα με τα οποία ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Έχουμε τις δημόσιες συμβάσεις, έχουμε τα δικαιώματα των επιβατών και έχουμε και την προσβασιμότητα. Uh, uh, Πρώτα απ' όλα, επειδή εδώ μιλάμε με, για δικαιώματα του ατόμου και έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους, η πτυχή της συμμετοχής είναι η πιο σημαντική. Πρωταρχική πτυχή που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη. Αυτό σημαίνει ότι όταν ορίζεται η προσβασιμότητα, αυτό θα πρέπει να ορίζεται σε όλους μας τους νόμους ότι οι διάφορες ομάδες ατόμων με αναπηρία θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις όταν ορίζονται οι προτεραιότητες, οι σπουδαιότητες και όταν ορίζεται τι ακριβώς σημαίνει προσβασιμότητα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είναι δύσκολο να δημιουργηθεί αυτή η δομή στη νομοθεσία μας, διότι δεν έχουμε σχεδιάσει τη νομοθεσία μας με αυτόν τον τρόπο. Για να ξεκινήσω από τις δημόσιες συμβάσεις. Πρώτα απ' όλα, Η ιδέα είναι ότι η υψηλή ποιότητα αγαθών και υπηρεσιών θα πρέπει να παρέχεται σε όλους τους πολίτες υπό καλές συνθήκες με καλή περιβαλλοντική ευθύνη και με φυσικά τις καλύτερες δυνατές τιμές. Όταν αγοράζουμε λοιπόν κάποια αγαθά, το ζήτημα είναι ότι εμείς ως άνθρωποι όταν χρησιμοποιούμε υπηρεσίες ε, διαφέρουμε μεταξύ μας. Πάντα θα πρέπει να να βλέπουμε τις διαδικασίες, τα, κατά τις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων, τις διάφορες ομάδες και τα διάφορα συμφέροντα. Όταν παρέχουμε λοιπόν υπηρεσίες στέγασης, υπηρεσίες πληροφορικής, είτε μιλάμε για επίσης δημόσιες μεταφορές, ιατρικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ταξί. Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες που παρέχονται, φορολογικές υπηρεσίες, θα πρέπει να συμβουλευόμαστε τους τελικούς χρήστες και ειδικότερα ενεργά να ε, απαιτούμε τη συμμετοχή διαφόρων ομάδων ατόμων. Σημαίνει αυτό ότι αυτές οι διαβουλεύσεις με τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς ε, και τους γενικότερους οργανισμούς που εργάζονται με τα άτομα αναπηρία θα πρέπει να συμμετέχουν, αλλά επίσης θα πρέπει δραστήρια να προσπαθούμε μέσω συνεντεύξεων, μέσω ερευνών ε, συμμετοχικής ε, συνεργασίας ε, μέσω γνωμοδοτήσεων θα πρέπει να προσπαθούμε να βλέπουμε πώς οι διάφοροι άντρες και γυναίκες με διαφορετικά είδη αναπηριών απαιτούν από τις υπηρεσίες τους και ότι ως άτομα τι θεωρούν θετική δράση για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας. Αυτό λοιπόν αλλάζει τις διαδικασίες σχεδιασμού και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων από τη σημερινή τους μορφή. Ουσιαστικά τις ανατρέπει. Ξεκινάμε δηλαδή από τους τελικούς χρήστες, τους ανθρώπους με διαφορετικές ανάγκες. Δεύτερον, και αυτό αφορά τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, τίθε το θέμα της επιτήρησης της ποιότητας των υπηρεσιών. Πολύ συχνά ένα άτομο, μια δημόσια υπηρεσία που αγοράζει μια υπηρεσία δεν τη χρησιμοποιεί το ίδιο. Το ερώτημα είναι λοιπόν ποιος έχει το δικαίωμα να εποπτεύει την ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πολλές διαφορετικές ομάδες. Αν σκεφτούμε άτομα με γνωσιακές δυσκολίες ε, ή δυσκολίες επικοινωνίας, δεν είναι πάντα τόσο εύκολο να γνωρίζουμε, να έχουμε υπόψη μας τα δικαιώματά σας, να γνωρίζουμε τι ακριβώς σας είχε υποσχεθεί κάποιος όσον αφορά την ποιότητα της υπηρεσίας και να γνωρίζουμε πώς ακριβώς μπορείτε να κάνετε μια απέτηση ποιότητα σε περίπτωση που η υπηρεσία δεν είναι αυτή που σας είχαν υποσχεθεί ή αυτή που απαιτείται βάσει των αναγκών του συγκεκριμένου ατόμου. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στην Επιτροπή λοιπόν. Ακόμα βρισκόμαστε σε φάση διαπραγματεύσεων με πολλά εκρεμή σημεία όσον αφορά την οδηγία για τι δημοσίε συμβάσει. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να έχουμε ένα κείμενο ε, σε κάποιο άρθρο όπου θα αναφέρεται ο ρόλος των οργανισμών που συνεργάζονται με άτομα με αναπηρίες για παράδειγμα ώστε να διαδραματίζουν το ρόλο εποπτών. Θα πρέπει να αναγνωρίζονται, θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επισκέπτονται στους τόπους όπου παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες, να κάνουν έρευνες μεταξύ των χρηστών των υπηρεσιών, να συγκεντρώνουν εμπειρίες και εφόσον χρειάζεται να υποβάλουν κάποιο αίτημα στον πάροχο ή στη δημόσια υπηρεσία που είναι αρμόδια για την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Πολύ σοβαρά σας λέω ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι να ενδυναμωθούν οι φωνές των χρηστών από διάφορες ομάδες ατόμων με αναπηρία. όχι μόνο λόγω των προβλημάτων επικοινωνίας, των περιορισμών επικοινωνίας. Πολύ συχνά έχουμε μικρές ομάδες και ορισμένες φορές ε, ο αριθμός των ατόμων είναι πολύ περιορισμένων και οι φωνές τους δεν ακούγονται τόσο εύκολα, δεν είναι τόσο οργανωμένη η επικοινωνία τους. Συνεπώς δεν μπορούν να επιτύχουν πολλά. Με αποτέλεσμα ή τα αποτελέσματα να μην είναι επαρκή. Τα τρία λοιπόν στοιχεία τα οποία προτείνονται όσον αφορά τις δημοσίες συμβάσεις και τη σχετική νομοθεσία είναι πρώτον Αυτή η στρατηγική για τις δημοσίες συμβάσεις ε, θα πρέπει να υποχρεωτικά να περιλαμβάνει την υποχρέωση για τους δημόσιους υπαλλήλους και για τους πολιτικούς να διεξάγουν ενεργές ακροάσεις ώστε να αναγνωρίσουν τις ανάγκες ε, των ομάδων χρηστών και να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε άτομα με αναπηρίες. ή σε άτομα με δικές ανάγκες. Το δεύτερο είναι αυτό που ανέφερα το δικαίωμα ενός οργανισμού. Παρακαλώ σε ένα λεπτό να τελειώσετε γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Και τέλος, ε, να υπάρχει το δικαίωμα ε, υποβολής και διεκπέρευση αυτών των ετοιμάτων. Αυτά ήθελα να αναφέρω για τι δημοσιοσυμβάσει και στη συνέχεια θα ήθελα να αναφέρω ότι η προσβασιμότητα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι μα. Τη συζητάμε και θα θέλαμε να έχουμε τα σχόλιά σα. Μετά από μια έρευνα τη Επιτροπή, ανακαλύψαμε ότι μόνο 10% των ιστοτόπων παροχή δημοσίων υπηρεσιών είναι εξοπλισμένε με υπηρεσίε πρόσβαση για άτομα με ειδικέ ανάγκε. Αυτό είναι μεγάλο ζήτημα. Ένα ζήτημα συνταγματικών δικαιωμάτων και επίσης και τα δικαιώματα των επιβατών είναι ένα ζήτημα στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση ώστε να εντοπίσουμε τις ανάγκες για υπηρεσίες από πόρτα σε πόρτα για τους επιβάτες με αναπηρία. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου για, το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σύρπα. Τώρα το λόγο έχει ο Πεκατόμινεν, ο οποίος είναι ταμεία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τα άτομα με αναπηρίες. Ευχαριστώ, πολύ, Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν πρέπει να μιλήσω ως ταμείας. Θα δούμε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Έχουμε αυτή τη στιγμή ακόμη πολλούς φραγμούς στο δρόμο των ατόμων με αναπηρία. Δεν τους επιτρέπουν να επαφολούνται τις ελεύθερες κυκλοφορίες. Για παραδείγμα, εμείς τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουμε μεγάλα εμπόδια στην πρόσβαση βασικών αγαθών και υπηρεσιών και δεν μπορούμε να επιφεληθούμε με τον ίδιο τρόπο που οποιοδήποτε άλλος Ευρωπαίος πολίτης μπορεί. ο οδηγός για τις ελευθερίες του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αναπηριών που δημοσιεύθηκε φέτος καταγράφει λεπτομερώς τις συνθήκες και τους διάφορους φραγμούς που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία. Επιπλέον, η κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη, η προσβασιμότητα ποικίλει σημαντικά και οδηγεί σε μια κατάσταση κατακαιρματισμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγμα το οποίο επίσης και επιπλέον υπονομεύει την ελευθερία κυκλοφορίας των πολιτών με αναπηρία. Τα ΑΜΕ έχουν το δικαίωμα της ε, ψήφου, το, εκλέγει, το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε σε ισότιμη βάση με τους λοιπού συμπολίτε του. Ωστόσο, πολλά εμπόδια, είτε υλικά είτε πολιτικά, μας κόβουν το δρόμο στη διαδικασία αυτή της πολιτικής συμμετοχής και επί παραδείγματι δεν μας επιτρέπουν να συμμετέχουμε επίσης όρις στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις δημοτικές αρχές, που είναι δικαιώματα αναγνωρισμένων στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Χρειάζεται λοιπόν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερα με την υιοθεσία μιας νομοθετικής πρότασης για την πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες και αναφέρομαι βέβαια στην πράξη και την προσβασιμότητα που περιλαμβάνει μια σαφή και εκτεταμένη περιγραφή, έναν ορισμό εκτεταμένο της προσβασιμότητας και ένα ευρύ φάσμα με τις προδιαγραφές της προβασιμότητας για συγκεκριμένους τομείς. Ορισμένοι μηχανισμοί κυρώσεων επίσης θα πρέπει να θεσπιστούν για να καταστεί δυνατόν να καταγράφεται και να αποκαθίσταται ενδεχόμενη ζημία εις βάρος αμαία σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την νομοθεσία για την προσβασιμότητα. Η υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή, επίσης, από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι επίση απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα και αυτό μέσα από τα διαφορετικά ταμεία και από την νομοθεσία για τις δημόσιες προμήθειες. Όσον αφορά την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο, το Φόρουμ για τις Αναπηρίες πιστεύει ότι η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, την ψηφία, για το ψηφιακό θεματολόγιο θα προσφέρει την συνεισφορά του με μια οδηγία φιλόδοξη και περιληπτική. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε και στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα ή στο τόπους με πρόσβασιμότητα για τα αμαία. Επίσης πρέπει να αποδειχθεί, να αποδειχθεί η στράτευση στις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την ελευθερία της κυκλοφορίας, η διακίνησης για κάθε πολίτη με αναπηρία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Πέκα. Πρέπει να σας πω ότι ήρθε ο κύριος Κλάουδιο Μοργάντη, αντιπρόεδρος της διακομματικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα άτομα με αναπηρίες. Θα μας βοηθήσει μάλιστα στο μέρος εκείνο το ανοιχτό που θα πάρετε εσείς το λόγο. Και σίγουρα θα με βοηθήσει πολύ και τον ευχαριστώ πολύ. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, θα ήθελα να ακούσουμε την Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι υπεύθυνη για την ψηφιακή ατζέντα, την κυρία Νέλη Κρούς, παρακαλώ. Και αυτό μέσα από μια μαγνητοσκόπηση που μας έχει στείλει. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα λειτουργήσει χωρίς πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πάρα πολύ να βρίσκομαι εκεί μαζί σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μοιραστώ μαζί σας καλά νέα. Ξέρετε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι αποκλείονται από πρόσβαση σε διάφορες ιστοσελίδες και άλλες υπηρεσίες online. Και γιατί? Γιατί εμείς αγνοούμε τις ανάγκες τους και τα ερωτήματά τους. Και όμως η λύση μπορεί να είναι τόσο απλή και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμά μου σήμερα. Το διαδίκτυο προσφέρει πάρα πολλά εργαλεία, μέσα, υπηρεσίε και ανοίγει νέες κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες. Είτε για την πρόσβαση στην ε, ηλεκτρονική κυβέρνηση, είτε μένοντας ε, και έχοντας επαφή με φίλους και συγγενείς, είτε έχοντας πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας ε, υγεία μέσω του διαδικτύου. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Δεν είναι κρίμα να αποκλείεται κανείς από αυτά. Γιατί, έχει προβλήματα στην όραση για άλλου λόγου και να μην μπορείς να χρησιμοποιείς τέτοια ιστοσελίδε στο διαδίκτυο. Και όμως 80 εκατομμύρια άνθρωποι περιορίζονται στην πρόσβαση αυτή. Πολύ συχνά υπάρχουν λύσεις. Υπάρχουν ιστοσελίδες που μπορεί κανείς εύκολα να έχει πρόσβαση σε αυτές ή να μπορεί να έχει επαφή μαζί τους. Αλλά δεν τα καταφέρνουμε όμως να προσφέρουμε αυτή την πρόσβαση και παρόλο που μερικές χώρες έχουν υιοθετήσει κανόνες, συχνά δεν φτάνουν αυτοί ή δεν είναι συνεκτικοί μεταξύ τους. Και πολλές φορές αυτοί που θέλουν να αναπτύξουν τέτοια μέσα διαπιστώνουν ότι υπάρχουν διαφορετικές προδιαγραφές στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Ε, λοιπόν, αυτό θέλω να αλλάξω, αυτό θέλω να διορθώσω και να βάλω τις κυβερνήσεις να αποτελέσουν το καλό παράδειγμα. Γι' αυτό λοιπόν και προτείνουμε οι ιστοσελίδε μα να είναι τέτοιε ώστε να έχουν εύκολα πρόσβαση τα άτομα με αναπηρίε από ολόκληρη την Ευρώπη. Είτε ψάχνετε με θέση απασχόληση, είτε θέλετε να βρείτε θέση σε ένα πανεπιστήμιο, είτε θέλετε ε, να κάνετε ένα ραντεβού με ένα γιατρό, οι προτάσει μα θα έχουν σαν αποτέλεσμα να μπορείτε αυτό να το κάνετε εύκολα. Αυτοί που φτιάχνουν τι ιστοσελίδε δηλαδή να λαμβάνουν υπόψη του τι δικέ σα ανάγκη. Έτσι εκατομμύρια άνθρωποι θα έχουν πιο εύκολα πρόσβαση σε όλες αυτές τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι διάφορες χώρες. Και έτσι θα υπάρχει επίσης ώρες πρόσβαση όλων. Βέβαια, ιδεοδός όλες οι ιστοσελίδες θα πρέπει να έχουν τέτοια διευκόλυνση και όχι μόνο εκείνες των κυβερνήσεων. Και ελπίζω ότι πράγματι μετά την πρωτοβουλία μας αυτή θα έρθει η στιγμή που όλες οι ιστοσελίδες θα διαθέτουν την ίδια εύκολη πρόσβαση για όλους. Και έτσι και οι προμηθευτές θα μπορούν εύκολα να προσφέρουν τα προϊόντα τους. Σήμερα κάνουμε το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Ελπίζω ότι όλοι έχετε τον ίδιο ενθουσιασμό όπως και εγώ για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Προσβλέπω λοιπόν στα αποτελέσματα της διάσκεψης αυτής. Ελπίζω να έχετε καρποφόρες εργασίες για το πώς θα εφαρμοστούν σωστά τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Τώρα θα μπούμε στην συζήτηση της Ολομέλειας και θα δώσω την προεδρία στον κύριο Μοργάντη, ο οποίος θα προεδρεύσει του τμήματος αυτού της διάσκεψής μας που έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις σας. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε Ζητώ συγγνώμη που δεν κατάφερα να συμμετέχω σε ολόκληρη την ημέρα αυτή τη συνάντηση, αλλά βρισκόμουν στην Ιταλία για δεσμεύσει ήδη ανηλυμένε. Μου κάνει μεγάλη χαρά που μπορώ να παρευρίσκομαι εδώ σε αυτή τη σύνοδο που σχετίζεται με την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρία. Ένα από τα θέματα, τα πιο σημαντικά για το οποίο και εγώ ο ίδιος ε, έχω συμμετάσχει προσωπικά στην ομάδα για τα άτομα με αναπηρία. Θέλω να δεσμευτώ τόσο για την Ευρώπη, αλλά κυρίως και για τη χώρα μου. Μου είπαν να είμαι και συνοπτικός, θα παραμείνω λοιπόν στα ουσιώδη. Θα ήθελα να σας αναφέρω και μία νίκη που κατάφερα στη χώρα μου. Το παράδειγμα του των αυτοκινήτων για τα άτομα με αναπηρία πριν από μερικούς μήνες στην Ιταλία. Ήμασταν μία από τις λίγες χώρες, ίσως η μόνη χώρα που δεν είχε έγκυρο ε, έγκυρη ετικέτα για τα αυτοκίνητα για πρόσβαση στους χώρους πάρκινγκ για τους αναπήρους. Όταν πηγαίναμε σε άλλες χώρες, όταν ένας ε, αναπήρος πήγαινε σε μια άλλη χώρα δεν γινόταν δεκτός ε, με το αυτοκίνητό του. Επιτέλους έπρεπε και η Ιταλία να συμμορφωθεί με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και η πόλη μου ήταν η πρώτη στην Ιταλία που το υλοποίησε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ είμαι προσωπικά υπερήφανος αφού προέρχομαι από την Πάδοβα την πόλη που πρώτη υιοθέτησε αυτό το, αυτό το σήμα. Γι' αυτό θα συνεχίσουμε να ευαισθητοποιούμε τον κόσμο για αυτά τα θέματα σε δύο πτυχές. Πρώτα απ' όλα στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη και θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε επίσης και τους πολίτες των δικών μας χωρών, περιοχών οι οποίοι θα πρέπει να έχουν συνείδηση των δικαιωμάτων τους, των δυνατοτήτων που μπορούν να υπάρχουν και από την Ευρώπη που συχνά και η Ιταλία θεωρεί μακρινή, απούσα, αλλά και που και σε αυτό το μέτωπο θα πρέπει να διαδραματίσει το ρόλο της με περισσότερες υποχρεώσεις και ευθύνες για το μέλλον. Είναι φυσιολογικό. Βρισκόμαστε στην Ευρώπη και έτσι θα εξαρτώμαστε όλο και περισσότερο από την Ευρώπη. Η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να επιτελέσει το έργο ευαισθητοποίησης της ε, δυνατότητας για όλους τους πολίτες να έχουν ίσα δικαιώματα. Ήθελα να ξαναευχαριστήσω εσάς για την παρουσία σας και δίνω το λόγο στην Βέρα Μπορβαλόφτ, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Good afternoon. My name is Vera. Καλημέρα σας, λέγομαι Βέρα. Εκπροσωπώ τα άτομα με εγκεφαλικές βλάβες και τις οικογένειές τους. Είναι ο εγκέφαλος το πιο σημαντικό, το πιο βασικό όργανο του ανθρωπίνου ε, οργανισμού που ελέγχει όλα τα εσωτερικά όργανα αλλά και, τους εξωτερ... και τις εξωτερικές δραστηριότητες. Στην Ευρώπη έχουμε πάνω από 2 εκατομμύρια πολίτες κάθε χρόνο που έχουν επιβιώσει μιας εγκεφαλικής βλάβης. Μεγάλος αριθμός λοιπόν αυτών παραμένουν στη ζωή με μια όμως επίκτητη εγκεφαλική βλάβη, ABI ονομάζεται στα αγγλικά, και πολλοί είναι οι νέοι οι οποίοι μαθαίνουν να ζουν με νέα όρια στις δυνατότητές τους, χωρίς όμως ε, καμιά ε, πρόσφορη ε, βοήθεια, χωρίς κατάλληλη βοήθεια, αναγκασμένοι να μένουν κλεισμένοι στο σπίτι και να ε, ζουν ε, τον ένα χρόνο μετά τον άλλο βλέποντα τη ζωή του να περνάει. Δεν μπορούν να είναι πραγματικοί πολίτε, δεν μπορούν ε, ούτε καν να είναι ορατοί μερικέ φορέ. αυτό λοιπόν είναι πολύ δύσκολο να το αντιληφθεί ο μέσο άνθρωπο, διότι έχουμε να κάνουμε με κεφαλικέ βλάβε οι οποίε κυρίω τι συνειδησιακέ λειτουργίε μπορούν να επηρεάσουν. Παραδείγματο τη δυνατότητα να βρει κανεί τον δρόμο για το σπίτι του, να επικοινωνήσει με του άλλου, δηλαδή την πολύ απλή καθημερινή ζωή. Ένα άτομο λοιπόν που πάσει από κεφαλική βλάβη λέγεται ότι μπορεί να, έχει άλλες, να βρίσκει άλλε τις λύσεις ή να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής του, εφόσον όμως του δοθεί η κατάλληλη υποστήριξη και η απεριόριστη χρονικά ε, πρόσβαση στην ε, νοσοκομιακή υπόθαλψη, πράγμα το οποίο όμως δεν συμβαίνει δυστυχώς στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν χώρες οι οποίες ούτε καν αναγνωρίζουν την ύπαρξη του προβλήματος αυτού. Άλλες το αναγνωρίζουν, αλλά λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν περιορίσει σημαντικά την εμπλοκή τους, την υποστήριξή τους ε, προς τα ε, άτομα που πάσχουν από κεφαλική βλάβη και τη δυνατότητα για αποκατάστασή τους. Ε, ενώ λοιπόν ενώ λοιπόν υπάρχει σημαντικό χάσμα ανάμεσα στα όσα προβλέπει η Σύμβαση των Εθνών και η πραγματικότητα, καλούμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει δράση έτσι ώστε τα άτομα με κεφαλική βλάβη να μην, με επίκτητη κεφαλική βλάβη, να μην παραμένουν στο σκοτάδι και να του δοθεί μια ευκαιρία να ξεφύγουν και από την κρίση και να ε, ζήσουν ω ενεργοί πολίτε για να ζουν και να είναι ενσωματωμένοι μέσα στι κοινωνίε. Ευχαριστούμε πολύ. Δίνω τώρα το λόγο στον Φιλίπ Σαζάλα, Γαλλικό Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρίες για ε, τα άτομα με, τέτοιε τέτοιες δυνατότητες για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο. Θα ήθελα να επιμείνω σε δύο σημεία που μου φαίνονται ουσιώδης σημασία και που δεν αναφέρθηκαν επαρκώς σήμερα το πρωί. Όλοι έχουμε καταλάβει πόσο ενδιαφέρον έχει η συνθήκη των ΗΠΑ και την ευημερία που μπορεί να προσδώσει στη ζωή των ατόμων με ειδικέ ανάγκε στην Ευρώπη, εφόσον εφαρμοστεί σωστά. Αλλά για να γίνει αυτό θα χρειαστεί να είναι δεσμευτική, να έχει την ισχύ νόμου. Εμείς ε, τα άτομα με αναπηρίες έχουμε την εντύπωση ότι ορισμένα κράτη απλά καθησύχασαν τη συνείδησή τους επικυρώνοντας τη συνθήκη των ε, Ηνωμένων Εθνών και πολύ γρήγορα κοιτούν να την παρακάμψουν ή και να μην την εφαρμόσουν. Έτσι λοιπόν μια απόφαση του Αρίου του της ε, προβλέπει ότι ορισμένα άρθρα τη συνθήκης δεν μπορούν να εφαρμοστούν στη χώρα μας γιατί δεν είναι επαρκώς ακριβή. Ουσιαστικά οι λόγοι είναι οικονομικοί οι οποίοι οδηγούν την κυβέρνησή μας ε, να μην ε, εφαρμόσει αυτή τη συνθήκη. Θέλουμε λοιπόν την ισχυρή στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να έχει νομοθετική, νομική ισχύ όπως όλοι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου. Είναι υπεράνω τη εθνική νομοθεσία και υποχρεώνουν τα κράτη που τις έχουν κυρώσει να τροποποιούν τους νόμους τους ανάλογα. Ένα από τα εμπόδια για την εφαρμογή αυτής της συνθήκη είναι ότι η κοινωνική νομοθεσία εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μέλων το οποίο αποτελεί ε, ε, φρένο για την εφαρμογή της συνθήκης. Όπως είπαν ορισμένοι ομιλητές σήμερα το πρωί, μια ενωμένη Ευρώπη δημοσιονομικά, κοινωνικά, θα επιτρέψει την καλύτερη εφαρμογή της συνθήκης. Θα θέλαμε να υπάρξει λοιπόν δέσμευση, θα θέλαμε όταν δεν εφαρμόζεται η συνθήκη αυτή να μπορούν να προσφύγουν κατάλληλα τα άτομα με αναπηρίες δικαστικά ώστε να αποτελεί υποχρέωση για τα κράτη που την έχουν κυρώσει. Ευχαριστώ πολύ. Υπολογίζουμε στη στήριξη της Ευρώπης για να γίνουν όλα αυτά στο μέλλον. Ευχαριστώ. Επόμενος είναι ο Χαροκόπο από την Ελληνική Ένωση για άτομα με αναπηρία. Έχετε δύο λεπτά. Thank you. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Πρόεδρε του EDF, κύριε και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, συνάδελφοι σα. Είναι για μένα ιδιαίτερη τιμή που παριστάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ω ένα από του αντιπροσώπους ελληνική εθνική ομοσπονδία ατόμων με αναπηρία. Η επερχόμενη υιοθέτηση μια ευρωπαϊκή πράξη προβρασιμότητα αποτελεί ορόσημο για την καθολική και ποιοτική αναβάθμιση του δοημένου και φυσικού περιβάλλοντο σε συνδυασμό με τη χρήση όλων των εφαρμογών τη σύγχρονη τεχνολογία. Στοχό είναι η διασφάλιση τη ισότητα, τη αυτονομία και τη ανεμπόδιση προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία η οποία στην ουσία αποτελεί πρόσβαση στην κοινωνία, εξίσωση ίσων ευκαιριών, συμμετοχή και εξάλληψη των διακρίσεων. Είναι υποχρέωσή μα να καταστήσουμε σαφέ ότι η ενίσχυση των διατάξεων για την προσβασιμότητα πρέπει να υποστηριχθεί από τι κυβερνήσει όλων των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα άθρα τη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τα δικαιώματα των ατόμων αναπηρία. Η Σύμβαση αποτελεί την πρώτη διεθνή ε, συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχει επικυρώσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση και καλύπτει αστικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα των ατόμων αναπηρία. Λαμβάνοντα υπόψη, υπόψη μα ότι τα άτομα αναπηρία και οι οικογένειέ του έχουν, έχουν πληγεί δραματικά από την παρούσα οικονομική κρίση και βιώνουν το πιο επώδυνο τρόπο την υποβάθμιση του δημόσιου συστήματο κοινωνική φροντίδα και εκπαίδευση πιστεύω ότι είναι επιτακτική ανάγκη να συστρατευτούμε υπό τη σκέψη του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων Απειρία ως πιο αντιπροσωπευτικό κίνημα. Εν μέσω κρίσιμων κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων καλούμαστε να συνιστήσουμε και να διεκδικήσουμε μια υφόρο κοινωνία αλλά και αλληλοσεβασμού. Θα επιθυμούσα τέλος να συμπληρώσω ότι η έννοια της η οποία έχει ταυτιστεί με τα άτομα αναπηρία στην πραγματικότητα μου. Η δυνατότητα δηλαδή να μπορεί κάθε άτομο αυτόνομα με ασφάλεια και άνεση να χρησιμοποιήσει υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά, αλλά επιπροσθέτως να επικοινωνεί και να πληροφορείται αποτελεί βασική παράμετρο που κατοχυρώνει θεμελιώδης δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης και επιλογής κάθε πολίτη της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Δίνω τώρα το λόγο στον Ζαν Λουξιμό, πρόεδρο του Disability People's International. Έχετε δύο λεπτά. Merci. Ευχαριστώ, κύριε πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι. Εδώ ε, κάνουμε τις συνεδρίες του Τρίτου Κοινοβουλίου των Ατόμων με Αναπηρία για να επιβεβαιώσουμε τα δικαιώματα και τον τρόπο με τον οποίο εμείς που έχουμε περιορισμένες δυνατότητες αντιμετωπίζουμε μια κρίση εδώ και πολύ καιρό, ίσως κρίση από την ημέρα που γεννηθήκαμε. Πώς μάθαμε όμως την κρίση αυτή να την ξεπερνούμε, να την αντιμετωπίζουμε και ίσως μερικές φορές και παρά την κρίση, την διαρκή κρίση που ε, ζούμε από τη μέρα που γεννηθήκαμε να βρίσκουμε τις λύσεις. Και αν υπάρχει ειδικό στις κρίσεις, αυτό είμαστε εμείς. Αν υπάρχει ειδικό στην εξέβρεση εναλλακτικών λύσεων, είμαστε εμείς. Και αν υπάρχει ανάγκη να ανεβρεθούν λύσεις και να αναζητηθούν τα, τα μυαλά εκείνα και οι εγκέφαλοι που μπορούν να, βρουν, να βοηθήσουν στην εξέβρεση λύσεων και στη έξοδο από την κρίση, αυτοί είμαστε εμείς. Εμείς που έχουμε μάθει να ξεπερνάμε τους φραγμούς, έχουμε την ικανότητα, έχουμε τη δεξιότητα και απαιτούμε τώρα να αξιοποιηθούμε και σαν μέσον για την ανάπτυξη του κοινού καλού. Μια πολιτική λοιπόν πραγματική συμμετοχής, μια συμμετοχή η οποία δεν θα είναι μόνο κατά το δοκούν, δεν θα ζητείτε μόνο κατά το δοκούν, ε, αλλά και που θα προχωρεί κατά τρόπο πλαισιωμένο και κατά τρόπο αμοιβόμενο, έτσι ώστε ο κάθε αμαία να έχει τη θέση του, να αξιοποιείται, να ε, την χάρη σεβασμού με τις ικανότητες του και να προσφέρει στο κοινό καλό. Χρειαζόμαστε κριτήρια που θα προσδιορίζουν αυτή τη συμμετοχή και την παρουσία μα στην Τράπεζα των Συζητήσεων και των Διαπραγματεύσεων, που όμω δεν αρκεί. Μπορεί να είναι απαραίτητο στοιχείο, αλλά δεν αρκεί να είμαστε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων. Χρειάζεται η συμμετοχή μα και να εξασφαλιστεί η παρουσία μα σε κάθε στάδιο τη ε, προόδου και τη εξέλιξη και της υλοποίηση νομοθεσία Πρέπει να είναι παραγωγική, δηλαδή σαφώ ε, περιγεγραμμένη ε, και προσδιορισμένη αυτή η συμμετοχή μας και με την αντίστοιχη δημοσιονομική στήριξη βεβαίω. Ευχαριστώ. Euh, euh, Ευχαριστώ πολύ. Όποιος λαμβάνει το λόγο παρακαλώ να μην ξεχνάει να σηκώνει το χέρι του για να τον βρίσκει η κάμερα. Μην το λησμονείτε. Ευχαριστώ. Jimmy Bowling. Jeremy Bolling, από την ανεξάρτητη, από την αυτόνομη ζωή. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι. Πολλοί είναι οι φραγμοί, άμεση και έμεση. Τους γνωρίζουμε πολύ καλά. Μιλάμε για προσβασιμότητα, για απουσία υπηρεσιών. Μιλούμε για σχέδια προσωπικής υποστήριξης, για περικοπές στα ερωτικά ταμεία. Οι επισκέψεις μου σε θεσμικά όργανα με έφεραν σε επαφή με ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσμενή κατάσταση ε, παρά τη θέλησή τους, ε, βρίσκονται ε, σε δεινή κατάσταση, κλαίνουν, παραπονιούνται, ζητούν να μπορούν να ζήσουν ανεξάρτητη ζωή, αλλά ενώ έχουν πολλές φορές την ενώ ζουν, έχουν πολλές φορές συνδιώκτη κατοικία, είναι υποχρεωμένοι να ζουν μέσα σε φύλακες και να μην έχουν ανεξάρτητη ζωή. Δεν μπορούν λοιπόν να ε, εξασφαλίσουν αυτό που χρειάζονται. Εμείς προσπαθούμε μέσα από, από τον ιστότοπό μας να βοηθήσουμε και να δείξουμε τι είδους, τι είδους μέσα χρειάζονται. Είχαμε παραδείγματι έναν ε, φοιτητή ο οποίος εξασφάλισε μια υποτροφία για να σπουδάσει, βούλγαρος στην Αυστρία, αλλά δεν μπορούσε να έχει άτομο συνοδείας μαζί και αναγκάστηκε να καταλήψει τις σπουδές. Αντίστοιχα μια άλλη κοπέλα με υποτροφία για διδακτορικό που αναγκάστηκε να καταλήψει. Άρα χρειάζονται Χρειάζεται ρεσιμότητα ω προ κάθε τύπου χρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ερευνητικά κονδύλια, παραδείγματι και χρηματοδότηση των προγραμμάτων των ερευνητικών ε, υπάρχουν πολλές δυσκολίες, πολλές φορές ε, δεν έχουμε καν κατάλληλο τρόπο για να συναντιόμαστε, δεν υπάρχει δηλαδή ξενοδοχείο με επαρκές συνθήκες προσβασιμότητας για τα αμαία ε, και είμαστε υποχρεωμένοι να παραμένουμε σε, σε μέρη τοποθεσίες άλλες που μας προσφέρουν στέγη μόνο και μόνο επειδή έχουν τις κατάλληλες συνθήκες πρόσβασης για μας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να ε, προωθηθεί το σχετικό ψήφισμα και οι ορισμοί. Πρέπει πλέον να τιμωρούνται αυτοί οι οποίοι ε, προβαίνουν σε, αυτά τα, σε αυτή την αδικία, γιατί μόνο έτσι θα μάθουν και δεν θα επαναλάβουν τις αδικίες στο μέλλον. Επόμενος ε, Λίβεν της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τον για το σπίνα μπίφιντα και τον αντροκεφαλισμό. Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου επιτρέπετε να μιλήσω εκ μέρους της ε, Διεθνούς Νομοσπονδίας για τους 200.000 ε, Ευρωπαίους που ζουν υπό τέτοιε συνθήκες και τις οικογένειές τους και να σας δώσω τη δική τους προοπτική σε αυτό το σημαντικό φόρουμ σε αυτό το έτος ενεργούς γύρασης και ελεγγύης μεταξύ των γενναίων και αναμένοντας το επόμενο έτος, το ευρωπαϊκό έτος για τους πολίτες, εμείς διερευνούμε την κατάσταση των των ανθρώπων με δυσχυδή ε, ράχη. Ε, αυτοί οι άνθρωποι με δύσκολη ράχη και υδροκεφαλία ε, αυτή η επεκτηνόμενη γυράσκουσα ομάδα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερους φραγμούς για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία. Αυτά οι φραγμοί οφείλονται στην έλλειψη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, απασχόληση, παιδεία, σημαντικές ανισότητες. Κοιτώντας αυτούς μαθαίνουμε για τις επόμενες γενιές. Το να επιληθεί αυτό το ζήτημα δεν είναι θέμα χρημάτων, είναι θέμα στάσης σε ένα εγγραφό που ονομάζεται Your Internal Investments οι αιώνες επενδύσεις σας είναι ε, έχουμε συμπεριλάβει έννοιε που θα πρέπει να καταλάβουν όσοι χαράσουν πολιτική. Το πρώτο πρέπει να κάνουν είναι να γνωρίσουν και όχι να αγνοούν την κατάσταση. Μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Τα παιδιά με δυσχύδη ράχη και υδροκεφαλία συνήθως έχουν ε, πρόσβαση σε φροντίδα ε, πολυμορφείς και όταν φτάσουν στην ηλικία των 21 δεν μπορούν πλέον να λάβουν αυτή την ε, φροντίδα από διάφορους ιατρικούς τομείς. Μόλις ε, αναγνωριστεί αυτή η δύσκολη κατάσταση μπορούμε να συνεργαστούμε με όσου χαράσουν πολιτικέ ώστε να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει και να διασφαλίσουμε ότι θα άρουμε του φραγμούς ενεργού συμμετοχή των πολιτών για ανθρώπου με δυσχεδία και υδροκεφαλία. Τώρα δίνω το λόγο στην Τερέζα Παραγιών, της Ισπανικής Επιτροπής Εκπροσώπων Ατόμων με ε, ε, δυσκολίες δανειτικές για δύο λεπτά. Ε, Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου που μπορώ έτσι ενεργά να συμμετάσχω στο σημερινό φόρουμ. Οι άντρες και οι γυναίκες με αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποφέρουμε από πρώτο χέρι τις ε, καταστροφικές συνέπειες της ευρωπαϊκής κρίσης που είναι μια κρίση όχι μόνο οικονομική, δημοσιονομική, είναι και κοινωνική. Στις 2 Δεκεμβρίου, για πρώτη φορά στην ιστορία του κινήματος, στη Μαδρίτη είχαμε πορεία των ατόμων με αναπηρίες. Έγινε μια διαδήλωση, μια πορεία που σύμφωνα με την αστυνομία συμμετείχαν πάνω από 90.000 άνθρωποι. 90.000 άνθρωποι το Φέρμι που εκπροσωπεί πάνω από 7.000 ενώσεις και πάνω από 4 εκατομμύρια πολίτες οργάνωσε την διαδήλωση αυτή, τις διαδηλώσεις αυτές, τις πορείες. Το θέμα της ισότητας, της ένδυας, του κοινωνικού αποκλεισμού είναι πράγματα που έχουν τα άτομα, αλλά πολύ πιο σημαντικά έχουν να κάνουν με την κοινωνική συνοχή. Αυτή πλήττεται. Χρειάζεται λοιπόν μία δράση. Η Φέρμη με την ΟΝΘΕ που είναι η οργάνωση των τυφλών της Ισπανίας τον Ιανουάριο που μας πέρασε έφτιαξαν μια πλατφόρμα για τον τριτογενή τομέα της ενεργούς δράσης. Μια πλατφόρμα η οποία αποτελείται από εκατοντάδες μειονότητες που εκπροσωπεί πάνω από 9 εκατομμύρια πολίτες, γυναίκες και άντρες. Είναι αναγκαίο να γίνονται επενδύσεις στον κοινωνικό τομέα, στο ανθρώπινο δυναμικό δηλαδή και στην κοινωνική συνοχή. Η καινοτομία σίγουρα παίζει καθοριστικό ρόλο. Όπως πολύ καλά το γνωρίζετε εσείς, οι κύριοι τομείς όπου δουλεύουμε στον κοινωνικό τομέα και στην καινοτομία είναι ακριβώς την απασχόληση. Απασχόληση για όλους, εκπαίδευση, ενημέρωση και κοινωνική ένταξη. Τα άτομα με αναπηρίες, ακριβώς σε αυτούς τους τομείς είναι η ομάδα εκείνη ανθρώπων που κινδυνεύει περισσότερο με αποκλεισμό. Και γι' αυτό ακριβώς σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Ευρώπης. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια των χωρών μελών. Σήμερα περισσότερο από ποτέ έχουμε ανάγκη από πολιτικές και από μέτρα τα οποία να μας προστατεύουν και να υποστηρίζουν τα δικαιώματά μας δικαιώματα που αγωνιστήκαμε τόσο για να κατακτήσουμε. Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε τη βοήθεια των Ευρωπαϊκών Κοινωνικών ε, Κονδυλίων. Ευχαριστώ πολύ. Από την Ισπανία περνάμε στη Σουηδία. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Λάρς Λίντμπεργκ της Σουηδικής Ομοσπονδίας Ατομών με Αναπηρία. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. He's not here. Δεν βρίσκεται εδώ. Το όνομα μου είναι Ράγνερ Βέρ και είμαι πρόεδρος ε, αναπληρωτής ε, του Λασινγκμπέργκ δεν μπορούσε να βρεθεί εδώ σήμερα το απόγευμα. Το θέμα που θα ήθελα να θέσω αφορά το γεγονός ότι εμείς εκπροσωπούμε 8 εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρη την Ευρώπη, ανθρώπους με αναπηρία και το ερώτημα είναι τι μπορούμε να επιτύχουμε. Εμείς είμαστε άνθρωποι με γνώσεις, με εμπειρία, με εμπειρογνωμοσύνη και θα ήθελα να ε, αναφερθώ στο κείμενο της Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών διότι μιλάει πολύ καθαρά εδώ αν κοιτάξετε στο άρθρο 4 στις γενικές δεσμεύσεις στο σημείο 3 αναφέρεται στη διαβούλευση και πιστεύω ότι κάθε θεσμικό όργανο και κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει εμάς ως εμπειρογνώμονες θα ήθελα να το τονίσω αυτό γιατί μιλάμε για ελευθερία κυκλοφορίας και ελευθερή άσκηση της ιδιότητας του πολίτη για άτομα με αναπηρίες. Θα πρέπει να άρουμε τους φραγμούς, τα προσκόμματα, η ελευθερία μετακινήσεις, κυκλοφορίας αποτελεί έναν από τους ε, ακρογωνίους λήθης της ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης. Ουσιαστικά αποτέλεσε προϋπόθεση που έθεσαν τα κράτη-μέλη, κυβερνήσεις. Πρέπει να κάνουν λοιπόν κάτι για την αντιμετώπιση των φραγμών προς την ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων με αναπηρία. Διότι όταν βλέπουμε φραγμούς για τους εργαζομένους, για ανθρώπους που θέλουν πρόσβαση σε παιδεία, αυτοί οι φραγμοί εμποδίζουν την ανάπτυξη της Ευρώπης και την διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να διδραματίσει σημαντικό ρόλο για την προώθηση αυξημένης, βελτιωμένης κινητικότητας για άτομα με αναπηρίες μέσω της ανάπτυξης της σχετικής τυποποίησης και ενίσχυσης των οδηγιών και των διαφορών δραστηριοτήτων που θα προωθήσουν ε, παιδεία για όλους. Εδώ μπορούμε να κοιτάξουμε για παράδειγμα το σχεδιασμό, μπορούμε να να ξεκινήσουμε πρωτοβουλίες σε αυτό το τομέα. Όσον αφορά τώρα την στρατηγική έρευνα και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και επενδύσεις στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να το προωθήσουμε και η Σιουδική Αντιπροσωπεία θα ήθελε ιδιαίτερα να τονίσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για την διεθνή τυποποίηση που θα πρέπει να χρησιμοποιεί ως βάση την παιδεία για όλους διότι για ένα διεθνές κίνημα για άτομα με αναπηρίες πρέπει να διασφαλίσουμε ότι μεριμνάμε επαρκώς για αυτά τα θέματα σε θέματα τυποποίησης η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εγγυηθεί ότι τα ευρωπαϊκά ταμεία έρευνα και τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να επιταχύνουν τι επενδύσει ώστε να προχωρήσουμε προ μια κοινωνία χωρί αποκλεισμού. Αυτό θα θέλαμε να προσαρτηθεί στα πρακτικά. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσετε τον λόγο. Τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Μπάνγκλιν Στέφαν Στότυρ, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοφών για τρία λεπτά. Καλησπέρα σας. Θα χρησιμοποιήσω την ε, νοηματική. Εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ένωση των Κοφών με ε, μέλη εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ορβηγία, την Ελβετία και την Ισλανδία. Έχουμε κάνει έρευνα σε όλη την Ευρώπη, τα κράτη-μέλη, για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και βλέπουμε ότι το 85% των ατόμων με αναπηρία είναι από ανθρώπους κοφούς ή που χρησιμοποιούν την ομαδική γλώσσα και καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι χρησιμοποιούνται πολύ οι διερμηνείς της νοηματικής. Ρωτούμε λοιπόν και βλέπουμε ότι 50% 50% ε, μας λένε ότι είναι πολύ χαμηλή η προσφορά διερμηνέων της νοηματικής ε, ή και μηδενική για μεγάλο ποσοστό των ε, κοφών ε, στην Ευρώπη. Άρα είναι πολύ περιορισμένη η χρήση της νοηματικής και ως εκ τούτου η ελευθερία διακυκλοφοριας που είναι πολύ σημαντική όμως για τους πολίτες μας και πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν την διερμηνία της νοηματικής. Αυτό σημαίνει εν ολίγης ότι αν θέλουμε να έχουμε την ελευθερία της κυκλοφορίας χρειάζεται να έχουμε και νομοθεσία εγκάρσια, σαφή, η οποία θα εξασφαλίζει την προσβασιμότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εθνικό επίπεδο στον τερμινέ της πνευματικής και ταυτόχρονα μια μορφή τυποποίησης για την κατάρτιση των ε, διερμηνέων της νοηματικής ανά την Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι εμείς ε, οι διερμηνείς της νοηματικής είμαστε 800 8.500 και έχουμε μόνο 6.000 διερμηνείς νοηματικής, ε, χρειαζόμαστε μια σεφέστερη νομοθεσία και ποιοτική κατάρτιση για τους διερμηνείς μας. Και έτσι θα μπορούμε όλοι να αξιοποιούμε την ελευθερία κυκλοφορίας, διακίνησης στην Ευρώπη. Δίνω το λόγο στην κυρία Λετήσια Πετιτζάνα, Γαλλικό ε, Συμβούλιο για άτομα με αναπηρίε. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Merci. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ως εκπρόσωπος νέων με αναπηρίες, θέλουμε να προσέξετε όλους ιδιαίτερα τις δικές μας ανάγκες και τις δικές μας προσδοκίες όσον αφορά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στον τομέα της εκπαίδευσης, για παράδειγμα, θα θέλαμε εγγύησεις να υπάρχει ισότητα με τους άλλους φοιτητές ή τους άλλους καταρτιζόμενους, να έχουμε την ίδια πρόσβαση λοιπόν στην κατάρτιση όπως γίνεται ακριβώς και με τους υπόλοιπους νέους. Η αλήθεια είναι ότι αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα στην κινητικότητά μας. Έτσι δεν μπορούμε να ταξιδέψουμε αρκετά, να σπουδάσουμε, να καταρτιστούμε για να προετοιμαστούμε για την αγορά εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα έπρεπε να διασφαλίσει την κοινωνική επίση συμμετοχή μας στην ψυχαγωγία, στον αθλητισμό, στα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη, εν πάση περιπτώσει. Μια πολιτική ένταξης σημαίνει ότι χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις που να λαμβάνουν υπόψη τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Είναι πολύ σημαντικό και με αυτό θα τελειώσω να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τον κοινωνικό διάλογο με τους νέους, η Ευρώπη δηλαδή με τους νέους, ώστε οι νέοι να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως την ε, ανάπτυξη και στην οικοδόμηση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής στην οποία να συμμετέχουν όλοι. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Μαρτίνα Άντερσον. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ τους οργανωτές που συγκέντρωσαν εδώ τόσο κόσμο με ένα τόσο ωραίο πρόγραμμα. Είναι κάτι που βλέπω όλο και περισσότερο στην Ιρλανδία, τη δική μου χώρα, ότι δηλαδή η κρίση χρησιμοποιείται σαν άλοθη, σαν πρόσχημα για να υπάρξουν όλο και περισσότερες περικοπές στην χρηματοδότηση που απευθύνεται σε άτομα με αναπηρίες. Στη Βόρεια Ιρλανδία το DLA έχει διαλυθεί περίπου. Έχει αλλάξει και το όνομα και έχουν μεταφερθεί πόροι. Και έτσι τελικά δεν μπορούν τα άτομα με αναπηρίες να ζουν με την αυτονομία που μπορούσαν να ζήσουν μέχρι τώρα. Όμως, ακριβώς τώρα που υπάρχει οικονομική κρίση, εμείς πρέπει να ενισχύσουμε τα άτομα που βρίσκονται στο περιθώριο, να τα προστατεύσουμε και όχι να υποστούν τις μεγαλύτερες περικοπές. Και αυτό θέλω να το πω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάποιος ήταν με αναπηρική καρέκλα και διαπίστωσα ότι στις Βρυξέλλες μόνο δύο εστιατόρια υπήρχαν τα οποία μπόρεσαν να επιτρέψουν την ε, πρόσβαση και στη τουαλέτα και στο εστιατόριο σε άτομα με αναπηρία με αναπηρική καρέκλα. Και είμαστε στην πρωτεύουσα της Ευρώπης. Εγώ νόμιζα ότι κάτι τέτοιο δεν θα το συναντούσα ποτέ. 2012 είμαστε, έτσι, όχι 1812. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε περισσότερες προσπάθειες ώστε να υπάρχει προσβασιμότητα για όλους. Τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να χαίρουν της ελευθερίας διακίνησης, κάτι που αναφέρεται στις συνθήκε και να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα, ο Νίρο Ζόλτα, Ουγγαρία από την Οργάνωση για Άτομα με Αναπηρίες. Τρία λεπτά παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, φίλοι, η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ηλικία, με το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν, ανάλογα με την κοινωνία στην οποία βρίσκονται και τον τρόπο με τον οποίο αυτή η κοινωνία μεταχειρίζεται τα άτομα με σε Αυτό είναι νομίζω ένα πολύ σημαντικό ε, μήνυμα για όποιον καλείται να χαράξει νομοθεσία για τα δικαιώματα για τα άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Σύμβασης των Εθνών. Και θα ήθελα να πω ότι όταν ήμουν δύο ετών έχασα την ακοή μου λόγω μιας υπερβολικής δόσης ε, στη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθούσα. Και βλέπω ότι έχει όπως και εγώ μεγαλώσει μια ολόκληρη γενναία που δεν είχε τη δυνατότητα να, χρησιμοποιήσει την νοηματική γλώσσα την ουγγρική και δεν γνώρισε, δεν είχε την αναγνώριση από τις αρχές των ιδιαίτερων αναγκών. οι επιλογές των κρατικών αρχών ήταν να επιβάλλουν στα άτομα με αυτή την ε, αναπηρία να ε, μιλήσουν σαν άνθρωποι χωρίς προβλήματα, να προσπαθήσουν δηλαδή να μάθουν να μιλούν. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με το προσδιορισμό της ζωής, της μοίρα, ολόκληρης της ζωής ενός ανθρώπου. Ένα παιδί λοιπόν το οποίο ε, μεγαλώνει χωρίς προβλήματα ακοής μπορεί να μάθει πλήρως τη γλώσσα του, τη μητρική. Είναι η βάση αυτό της εκπαίδευσής του, της ανάπτυξής του κτλ. Όμως αυτό δεν συμβαίνει σε ανθρώπους όπως εγώ. Τα παιδιά που γεννιούνται με κόφωση, που δεν μπορούν να ακούσουν, μια και η μητρική μας γλώσσα δεν είναι η γλώσσα της μητέρας μας. Εμείς, άνθρωποι όπως εγώ, μάθαμε μία γλώσσα στα κρυφά. Στα κρυφά για να μπορέσουμε να καταστούμε μέλος μιας κοινότητας επικοινωνίας που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας. Γι' αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία για μας αυτή η σύμβαση, διότι λέει ότι πρέπει να προάγεται η διδασκαλία και μάθηση της νοηματικής γλώσσας και ότι πρέπει να υποστηρίζεται η γλωσσική ταυτότητα των ανθρώπων με προβλήματα ακοής. Πολλοί νόμοι έχουν ε, τεθεί σε ισχύ, θεσπίζοντας ένα νομικό πλαίσιο ή νομικό περιβάλλον. Έχουμε νόμους λοιπόν για ίσες ευκαιρίες, έχουμε νόμους για την εκπαίδευση. Για τις νέες όμως εκπαιδευτικές δραστηριότητες χρόνος δεν προσφέρεται. Αυτό που βλέπουμε είναι χωριστά εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία καλούνται να ε, ε, επιφορτιστούν με νέα καθήκοντα, ανάλογα με τη νέα νομοθεσία, να παρακολουθήσουν νέα προγράμματα χωρί απαραίτητα την κατάλληλη χρηματοδότηση. Πρέπει δηλαδή να του χορηγηθούν και τα κατάλληλα οικονομικά μέσα. Και ακόμη περισσότερο. Χρειάζονται υπηρεσίε διερμηνίας σιγά σιγά αυξάνεται ο αριθμό των προγραμμάτων στην τηλεόραση παραδείγματι που μεταδίδονται με παράλληλη διερμηνία στην νοηματική. Χρειάζονται όμω και ευκαιρίε ίσες σε κάθε επίπεδο τη ζωή για τα παιδιά και του άτομα με αναπηρία. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο σε όλη την Ευρώπη και πρέπει να βρούμε εκείνους τους συνταξιδιώτες που θα πορευτούν μαζί μας και που θα μας στηρίξουν στις προσπαθίες μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενη ομιλήτρια, Κορίν Κλέμοντ, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας της Αυτόνομης Εκπροσώπησης, για τέσσερα λεπτά. Bonjour. Je Καλημέρα, ονομάζομαι Κορίν Κλερμόν, προέρχομαι από τη Γαλλία. Σήμερα εκπροσωπώ την Εύσοδο. Η ΕΠΣΑ είναι η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα των Αυτόνομων Εκπροσώπων. Πρόκειται για άτομα με αναπηρία πνευματικά που μιλούν για τα δικαιώματά τους και τις ανάγκες τους. Η ιδιότητα του πολίτη στην Ευρώπη είναι για παράδειγμα το να ψηφίζει κανείς στις ευρωεκλογέ. Όλα τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να έχουν το δικαίωμα ψήφου. Οι εκλογές πρέπει να παρέχουν πρόσβαση. Αυτό δεν σημαίνει μόνο προσβασιμότητα στα ε, εκλογικά κέντρα. Είναι σημαντικό το πρόγραμμα των πολιτικών κομμάτων να είναι προσπελάσιμο σε όλους. Πρέπει να είναι ευκολονόητο. Χρειάζεται επίσης ενημέρωση για όλες τις εκλογές, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε σε τι χρησιμεύουν. Είμαστε πολίτες εξ ολοκλήρου. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να ενημερωνόμαστε, ώστε να μπορούμε να εκπληρώνουμε τα καθήκοντά μας ως πολίτες. Πρέπει επίσης να βοηθάμε τα άτομα με αναπηρίες για να θέτουν υποψηφιότητα σε εκλογές. Διότι ναι, γιατί να μην υπάρχει ένα άτομο με διανοητικά ε, ζητήματα ως μέλος του Ευρωκοινοβουλίου. Υπάρχει και ένα έγγραφο σε σχέση με τις ε, εκλογές για άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη. Καλό θα ήταν να αφιερώσουν πέντε λεπτά από το χρόνο τους οι ευρωβουλευτές για να το διαβάσουν και να συναντήσουν τους αυτόνομους εκπροσώπους. Αυτό θα μας έκανε να κερδίσουμε πολλά σε θέματα προσβασιμότητας. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Δίνω το λόγο στην κυρία Ιζαμπέλ Μπαγιώνα Στεμπαέρα, Ισπανική Επιτροπή Εκπροσώπων Ατόμων με Αναπηρίες. Έχετε δύο λεπτά. Αξιότιμοι συνάδελφοι. Το Προήμιο της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η οικογένεια, άντρες και γυναίκες που αναλαμβάνουν να φροντίσουν μια οικογένεια. Εγώ είμαι από αυτές τις μητέρες που τα άφησαν όλα για να φροντίσουν ψυχήτη και σώματι τον γιο μου αυτιστικό. Κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει τα άτομα με αναπηρίες άμα έχει περάσει από κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και τις οικογένειες. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε τη στήριξή μας στις οικογένειες, οι και να φροντίσουμε για την κοινωνική προστασία, την κοινωνική ασφάλιση, υπηρεσίες υγείας, ποιότητας, πρόσβαση στην κατοικία και αξιοπρεπή ζωή. Θέλουμε και αναγνώριση για αυτούς οι οποίοι έχουν αφιερώσει τα πάντα στη ζωή τους για να φροντίσουν κάποιο άτομο με αναπηρίες. Οι κυβερνήσεις πρέπει να καταλαβαίνουν ότι εμείς οι οικογένειες προσφέρουμε τέτοιες υπηρεσίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια και ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα όπως οποιοδήποτε άλλος πολίτης. Δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις, αλλά να επιτρέπεται η ένταξη των ατόμων αυτών στην κοινωνία και να έχουν και το σεβασμό μας. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο στην κυρία Βαράτη Σιμών Σουσάν, ε, Ουγγρική Ένωση για άτομα με αναπηρίε, για δύο λεπτά. Σα ευχαριστώ πολύ. Εκπροσωπώ την Ουγγρική Οργάνωση Βαρικών και Κοφών και θα ήθελα να πω ότι στην Ουγγαρία. Έχουμε με την έννοια ε, φραγμό ε, αναγνωρίζεται μόνο ο φυσικός φραγμός, ε, ο υλικός φραγμός δηλαδή στην προσβασιμότητα. Εδώ νομίζουμε λοιπόν θα πρέπει να αναγνωριστεί η δυνατότητα να καταρριφθούν όλοι αυτοί οι φραγμοί και τα εμπόδια και στην επικοινωνία και ιδιαίτερα για τους ε, βαρικούς οικοφούς πρέπει να εξασφαλιστεί μια αξιοπρεπής καθημερινή διαβίωση και δυνατότητα πρόσβαση στην ε, επικοινωνία. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι να μπορούμε να χρησιμοποιούμε την ε, νοηματική γλώσσα. Υπάρχουν διάφορες επίσης τεχνολογίες βίντεο που επιτρέπουν αυτή την ε, ιδιαιτερότητα, τη βελτίωση της κατάστασης και της καθημερινής μας ζωής. Είχαμε στην Ουγγαρία μία πρόσκληση έναν διαγωνισμό που θα μπορούσε να βελτιώσει την προσβασιμότητα σε τεχνολογία βίντεο για τα άτομα με προβλήματα ακοής, περικοή ή κόφωση και την πρόσβαση στη διερμηνία. Πιστεύουμε ότι μπορούν, εφόσον προσφερθεί αυτή η οικονομική βοήθεια, ιδιαίτερα η οικονομική βοήθεια για τα άτομα με προβλήματα ακοή ε, από την κυβέρνηση, θα μπορούν να συμμετάσχουν πλήρω στον επαγγελματικό βίο ε, και να συμμετέχουν στην κοινωνία. Υπάρχουν διάφορα μέσα στήριξης, υποστήριξης, βοήθειας, όπως και η ανάγνωση ε, των χιλέων όσον σημείο αναγνώρισης της ομιλίας, αλλά και πολλά άλλα μέσα που θα πρέπει να ε, μας βοηθήσει η κυβέρνηση να εξασφαλίσουμε. Δίνω το λόγο στον Ζωζέ Μανουελ Γκονζάλες για δύο λεπτά. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε. Θέλω να σας μιλήσω για κάτι που πιστεύω ότι είναι σημαντικό. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μιλάμε για την ισότητα, για την κατάργηση των εμποδίων. Όμως τα μέσα ενημέρωσης τι ρόλο παίζουν σε όλα αυτά. Η υπευθυνότητα των μέσων ενημέρωσης έχει μεγάλη σημασία, γιατί πρώτα απ' όλα ε, μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση όλοι οι πολίτες. Έπειτα, τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να ενθαρρυνθούν να προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρίες. Τρίτον, η κοινωνία πρέπει να καταλάβει μέσα από τα μέσα ενημέρωση, βέβαια, την πραγματικότητα που ζουν τα άτομα με αναπηρία στην Ευρώπη. Και τέταρτον, πρέπει να χρησιμοποιείται αυτή η γλώσσα τόσο σημαντική για όλου. Αλλιώ τα άτομα με αναπηρίε δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν ποτέ ολοκληρωτικά στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ε, ε, Τώρα Έχουμε ένα βίντεο του κυρίου Βαν Ρομπέη. Παρακαλώ τους τεχνικούς. The third European Parliament Καλωσορίζω τις εργασίες του Τρίτου Κοινοβουλίου των Ατόμων με Αναπαρία σήμερα. Με μεγάλη χαρά όμως δεν θέλω να σας απευθύνω και ένα μήνυμα με, αυτή την, ε, με αυτό το βίντεο ότι δηλαδή η διάσκεψή σα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για συνάντηση μεταξύ ανθρώπων με αναπηρία, με αναπηρία από ολόκληρη την Ευρώπη, προαγωγή του ενεργού διαλόγου και μια επικοδομητικής εταιρική σχέση, όπω έγινε και με τα προηγούμενα δύο κοινοβούλια. Η τρέχουσα διάσκεψη μπορεί να έχει πάρα πολύ σημαντικό αντίκτυπο στην πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα άτομα με αναπηρία. Πέρυσι έλαβα μέρο και εγώ στην ε, ομιλία για την κατάσταση τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, νόπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον Πρόεδρο τη Επιτροπή κ. Βαρόσο και τοποθετή αναφέρθηκα και στο θέμα αυτό και βλέπουμε σήμερα ότι η διάσκεψη σα αποτελεί μια συγκεκριμενοποίηση των όσων ε, είχαν υποθέσει εκείνη τη συνεδρίαση. Σήμερα λοιπόν κάνετε ει βάθο συζητήσει για τι τωρινέ και μελλοντικέ πολιτικέ για τι αναπηρίε στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ιδιαίτερα θα επικεντρωθείτε στη σημασία και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη των κατάλληλων πολιτικών και μέσων. Μαζί με τη Σύμβαση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αποδείξει τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών και μέτρων για τα άτομα με αναπηρία. Η πρώτη σχετική έκθεση, η έκθεση δηλαδή για την υλοποίηση της ε, σύμβασης που θα ε, ελέγξει η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αποτελεί ένα σημαντικό βήμα, καθοδηγεί τι μελλοντικέ δράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίε και κύριοι, σε μια στιγμή μεγάλων οικονομικών προκλήσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσκολλημένη στην αρχή τη προστασία των πιο ευάλωτων, των νέων, των γυναικών, των ατόμων με αναπηρία. Η δράσεις μας για την αποκατάσταση της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας έχουν ιδιαίτερο στόχο την προστασία και την διαφύλαξη του κοινωνικού κράτους, ε, της ε, κοινωνικής πρόνοιας, του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου δηλαδή, των ανθρώπων της Ευρώπης που είναι η ψυχή και η καρδιά της Ευρώπης μας. Σας ευχαριστώ και καλή επιτυχία σε εργασία σας σήμερα. Τώρα θα καλέσω εδώ στα έδρανα της Προεδρίας την Σισίλια Βινστρόμ, αντιπρόεδρο της Διακομματικής Ομάδας για τα άτομα με αναπηρίες, συναδελφό μου και θα καλέσω επίσης και τον πρόεδρό μας της Διακομματικής Ομάδας, Κώσα, εδώ στη θέση της Προεδρίας. Δύση. Καλησπέρα και από μένα, κυρίε και κύριοι. Είμαι η Σεσίλια Βίλστρομ. Είμαι ευρωβουλευτή από το 2009 εδώ και είμαι και αντιπρόεδρο της διακομματικής ομάδας για τα δικαιώματα των αναπήρων, όπου ο συναδερφός μου, εδώ ο Άνταμ, είναι ο πρόεδρος. Δεν βλέπω τη συνδική προσωπία, μα πού είσαστε. Α, δύο μόνο. Α, εντάξει. Τώρα βλέπω ότι υπάρχουν τόσοι Σουηδοί φίλοι εδώ μαζί μας σήμερα. Τώρα πέρα από τους Σουηδούς βλέπω Έλληνες, παντού Έλληνες βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και σας καλωσορίσατε όλοι οι Έλληνες, λέει στα ελληνικά η κυρία Ελπίζω να περάσετε μια μέρα με καρποφόρες εργασίες εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τότε που είμαι εγώ ευρωβουλευτής, πριν από τρία χρόνια δηλαδή, ήμουνα πριν 7 χρόνια στο Σουηδικό Κοινοβούλιο, έτσι. Όπως σας είπα, είμαι αντιπρόεδρος στη διακομματική ομάδα για τα άτομα με αναπηρίες και ειλικρινά θαυμάζω τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι τώρα. Έχουμε συνεργαστεί βέβαια με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τα άτομα με αναπηρίες που, είναι, που έχουν λάβει τόσο μεγάλη υποχρέωση υπέρ των ατόμων αυτών και του θαυμάζω ειλικρινά. Υπάρχουν τόσα πολλά θέματα και βέβαια δεν μπορούμε όλοι να τα κάνουμε όλα. Εγώ πάντως έχω ασχοληθεί με το θέμα της αυτονομίας στη διαβίωση. Και χαίρομαι που είμαι Σουηδή και περήφανη συγχρόνως που είμαι Σουηδή γιατί η Σουηδία είναι η μόνη χώρα στον κόσμο όπου η προσωπική βοήθεια για αυτονομία των ατόμων με αναπηρία είναι ένα δικαίωμα. Δεν κάνουμε καμιά διαφορά. 40% των ατόμων που χρησιμοποιούν αυτή την ατομική βοήθεια στη Σουηδία έχουν διανοητική καθυστέρηση. Πριν από μερικές εβδομάδες, ένα μήνα νομίζω, οργάνωσε ένα σεμινάριο εδώ για το πώς θα σταματήσει η ιδρυματοποίηση που ισχύει τόσο πολύ στην Ευρώπη. Σήμερα στην Ευρώπη μόνο η Νορβηγία και η Σουηδία έχουν καταφέρει να καταργήσουν τα μεγάλα ιδρύματα. Για να κλείσουν όμως τα ιδρύματα και στις άλλες χώρες πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και πρέπει οι κοινωνίες να προσφέρουν διαφορετικού είδους στήριξη. Δεν λέω ότι υπάρχει μία λύση που να κάνει για όλους, όχι. Η προσωπική λοιπόν αυτή αρρωγή είναι για τους περισσότερους ανθρώπους η μόνη δυνατότητα προκειμένου να μπορέσουν να αποφασίσουν οι ίδιοι για τη ζωή τους. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουν να ζήσουν με αυτονομία. Τώρα δεν ξέρω αν σας αρέσουν οι μοντέρνες ταινίες, οι καινούργιες, αλλά εγώ είδα μία πριν από λίγες εβδομάδες μόνο. Μία ταινία που αναφερόταν σε αυτό ακριβώς ε, το θέμα, την ε, διαβίωση με αυτονομία. Λέγεται του Σάμπλ. Σας Untouchables. Αν ε, έχετε την ευκαιρία, δείτε την. Είναι μια εξαιρετική ταινία και σημαίνει πολλά για τους νέους. Θα ήταν πολύ καλό να περάσει το μήνυμα της ταινίας αυτής τους νέους. Τώρα πέρα από αυτό, ο τίτλος της σημερινή μας συνάντησης είναι «Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες μέσα σε μια περίοδο κρίσης». Δεν είναι μυστικό βέβαια ότι σε περίοδους οικονομικών δυσκολιών οι πιο ευάλωτοι από τους ευάλωτους είναι αυτοί που πλήττονται και περισσότερο. Είναι αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο με το χειρότερο τρόπο. Γι' αυτό και οι υποχρεώσεις μας πρέπει να παραμένουν υποχρεώσεις, ακόμα και σε περίοδους κρίσης. Σε περίοδο παχαίων αγελάδων και ισχνών αγελάδων υποχρέωση είναι υποχρέωση. Γι' αυτό λοιπόν ιδιαίτερα σε δύσκολους καιρούς πρέπει να διασφαλίζουμε ότι κανένας δεν μένει χωρίς φροντίδα, κανένας δεν πρέπει να μένει πίσω. Αυτό βέβαια είναι πιο εύκολο να το πει κανείς παρά να το κάνει. Αλλά ήδη αν μπαίνει το πρόβλημα αυτό πάνω-πάνω στην ημερήσια διάταξη, όπως το κάνουμε σήμερα, και αν υπογραμμίσουμε και δείξουμε στον κόσμο ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες αν αγνοήσουμε αυτή την προτεραιότητα, τότε οι θύνοντες και όσοι παίρνουν τις αποφάσεις δεν θα μπορέσουν να παραβλέψουν το πρόβλημα. Εγώ προσωπικά χαίρομαι πολύ όταν ακούω το σλόγγαν αυτό «Να μην γίνει τίποτα για μας χωρίς εμάς». Πολύ καλό σλόγγαν αυτό, φαντάζομαι ότι το έχετε μάθει όλοι τώρα. Και ξέρω ότι πολλοί από εσά τα καταφέρνετε πάρα πολύ καλά. Τίποτα για μας χωρίς εμάς. Εσείς είσαστε ειδικοί. Εσείς γνωρίζετε καλά αυτά τα θέματα, τα θέματα σας. Και εγώ ως πολιτικός έχω την υποχρέωση, αλλά αποτελείτε κι εσείς έμπνευση για μένα όταν σας ακούω. Έχω την υποχρέωση λοιπόν να σας ακούω. Εμπνέομαι από αυτά που λέτε και λαμβάνω υπόψη μου τα όσα λέτε κάθε φορά που καλούμε να πάρω ε, πολιτικές αποφάσεις ή να νομοθετήσω. Να συνεχίσετε να μοιράζεστε τις ιδέες σας, τις εμπειρίες σας μαζί μας. Γιατί να ξέρετε ότι υπάρχουν πολλοί που σας ακούνε. Τα πράγματα έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν χωρίς εσάς. Και αυτό το λέω από βάθος καρδίας να έρχεστε να μας μιλάτε, ακόμα και να μας ενοχλείτε με τις ιδέες σας. Αλλά μην σταματήσετε ποτέ την επικοινωνία μαζί μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. And now I am happy to give... Και τώρα, με ιδιαίτερη χαρά, θα δώσω το λόγο στον κύριο Βαρδακαστάνη εκείνος θα ηγηθεί τη ψηφοφορία. Thank you. Thank you very much. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καταρχάς για τις πολύ σημαντικές τοποθετήσει σας. Προσβλέπουμε σε μια πιο στεναρή και πιο επικοδομητική ε, εταιρική σχέση με, με όλους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό το λέω τονίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του καλά καλά, ήταν ε, όχι μόνο ο πιο ισχυρός μας σύμμαχος, αλλά και ο πιο αξιόπιστος. Η ψηφοφορία λοιπόν τώρα. Ήταν πολύ εύκολη. γιατί όπως εξήγησε ο Πατ Κλάρκ το πρωί, θα ε, δείτε το κείμενο, έχουμε κάνει τις διαβουλεύσεις μας. Λαμβάνετε λοιπόν το κείμενο, προσπαθήσαμε να ενσωματώσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό όλα τα σχόλια που κατατέθηκαν και αυτό που μου μένει είναι να σας ζητήσω εάν δέχεστε αν εγκρίνεται το κείμενο του ψηφίσματός μας και ξεκινώ ερωτώντας αν είναι κανείς κατά του κειμένου ψηφίσματος, του σχεδίου ψηφίσματος που συζητούμε τον τελευταίο περίπου μήνα. Είναι κανείς κατά, παρακαλώ να σηκώσει το χέρι του. Όχι, είναι ξεκάθαρο ότι κανείς δεν έχει σηκώσει χέρι. Βλέπω πολύ καλά όπως ξέρετε. Και ο Γιάλος νομίζω ο φίλος θα ακούσει και όλα τις αντιρρήσεις. Καλώς, αποχές. Ουδής τέλεια και ως εκ τούτου το ψήφισμα εγκρίνεται ομόφωνα. Δεν δεν πρόκειται μόνο για ένα ψήφισμα. Τα όργανα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Αναπηριών σε συνεργασία και με τα μέλη μας αλλά και σε διαβουλεύσεις πρόκειται να ετοιμάσουν ένα προσωπικό σχέδιο με στόχο την ουσιαστική υλοποίηση του ψηφίσματος ώστε να αποφέρει καρπούς. Και είναι καθήκον των πάντων μας σήμερα που θα επιστρέψουμε στις πατρίδες μας, στις οργανώσεις μας, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αξιοποιήσουμε αυτό το κείμενο, αυτό το ψήφισμα σε κάθε επίπεδο, παντού, γιατί και εμείς χρειαζόμαστε να υπάρχει η απόδοση αυτού του ψηφίσματος, να φέρει αποτελέσματα αυτό το ψήφισμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς. The resolution... Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα. Ανυπομονώ να το δω, να το διαβάσω και να το κατανοήσω. Τώρα Φτάνουμε στις ε, δηλώσεις του Άνταμ Κώστα, του Προέδρου της Διακομματικής Ομάδας για τα άτομα με αναπηρίες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συμμετέχοντες, σήμερα δουλέψαμε σκληρά ολόκληρη την ημέρα. Πιστεύω ότι ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμπειρία και ένα πολύ ωραίο συνέστημα που ένιωσα που βρεθήκαμε εδώ εκπρόσωποι 500 ανθρώπων, 500 εκπρόσωποι ανθρώπων με αναπηρίες. Θέλω εδώ να σας πω ότι εκτίμησα πάρα πολύ τις εμπειρίες σας, τα όσα είπατε. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι καταφέραμε να βάλουμε και τις σκέψεις μας στο χαρτί. Θα ήθελα να συνοψίσω λιγάκι σε αυτά τα λεφτά που έχω στη διάθεσή μου τα πιο σημαντικά για μένα συμπεράσματα των σημερινών μας εργασιών. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι ότι το Ευρω... ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ίδιος, ήταν σαφής, αποφασισμένος. Φάνηκε αυτό από αυτά που μας είπε σήμερα το πρωί κατά την ε, κήρυξη της έναρξης των ε, εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ατόμων με Αναπηρίες. Αυτό που ακούσαμε σήμερα είναι ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι ζουν δυστυχώς κάτω από τα όρια της ε, Ένδιας και ότι μέσα σε αυτούς υπάρχουν όλο και μεγαλύτερα ποσοστά ατόμων με αναπηρίες. Θέλουμε να δούμε τι θα γίνει με την νομοθεσία ε, την επόμενη περίοδο. Τι θα αλλάξει στις πολιτικές δεδομένου ότι εξελίξει είναι αυτές που είναι. Τι θα γίνει και με τις δημόσιες συμβάσεις. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά την κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες και να προσπαθήσουμε να εκπονήσουμε νομοθεσία υπέρ τους. Αυτό ήταν το ένα. Κάτι άλλο ήταν ότι στις, ε, στην νομοθεσία πρέπει να διασφαλίσουμε και ότι προβλέπονται δεσμευτικά μέτρα, δεσμευτικά για να πετύχουμε πραγματικά τους στόχους μας. Επίσης, ο πρόεδρος Βαρδακαστάνης, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για άτομα με αναπηρίες, αναφέρθηκε σε δύο σημαντικά θέματα που θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω, γιατί νομίζω ήταν πολύ σημαντικά. είπε ότι οι παλιές συνταγές, οι παλιές λύσεις δεν λειτουργούν πια. Χρειαζόμαστε νέες τεχνολογίες, χρειαζόμαστε νέους τρόπους οργάνωσης της συνεργασίας μας, νέες λύσεις. Και είναι αλήθεια αυτό. Ο καθένας από μας το γνωρίζει αυτό. Ο καθένας από μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στη διακομματική μας ομάδα Περιμένουμε νέα νομοθετικά μέτρα για να διασφαλίσουν την ε, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες. Η ανάγκη είναι ιδιαίτερα αισθητή. Τώρα στη συζήτηση που ακολούθησε ακούσαμε εξαίρετες ιδέες και εξαιρετικά σχόλια. Φυσικά δεν έχω χρόνο τώρα να τα να επαναλάβω όλα, αλλά νομίζω ότι κάποια από αυτά πρέπει να τα υπογραμμίσουμε. Κάτι πολύ σημαντικό που άκουσα και που θα το λάβει υπόψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην νομοθετική μας δουλειά, στο νομοθετικό μας έργο. Γιατί αλλιώ οι νομοθετικές μας πράξεις δεν θα έχουν αξιοπιστία. Επίσης πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία σε διάφορα σημεία όπως είναι η απασχόληση, η εκπαίδευση και η προσβασιμότητα σε διάφορες υπηρεσίες. Αυτά τα ακούσαμε και τα έχουμε υπογραμμίσει ξανά και ξανά και είπαμε ότι το τομή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική ακριβώς ώστε τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία. Μιλήσαμε βέβαια και για την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρίες. Και είπαμε πόσο σημαντικό είναι η σύμβαση αυτή να τεθεί σε εφαρμογή τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της, όσο και στην κάθε χώρα μέλος χωριστά. Εν κατακλείδη. Θέλω να υπογραμμίσω και κάποια σημεία που ακούστηκαν για το μελλοντικό μας έργο. Πώς δηλαδή μπορούμε να προχωρήσουμε πιο πέρα και σε επίπεδο χωρών μελών. Η πρώτη βασική μας αρχή είναι ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία όταν έχουμε να κάνουμε με άτομα με αναπηρίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στις διάφορες οδηγίες, εκείνη για παράδειγμα για τα δικαιώματα των επιβατών, αλλά και σε άλλες οδηγίες, να υπάρχει συνοχή, ομοιομορφία και να καταλήγουμε σε εναρμόνιση να ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με άτομα με αναπηρίες, τα οποία τα αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Επίσης, αναφερθήκαμε και στην κατάσταση των γυναικών με αναπηρίες. Είπαμε ε, επίσης ότι υπάρχουν γυναίκες θύματα εγκληματικών πράξεων που είναι δύο φορές θύματα. Αναφερθήκαμε επίσης στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και ότι πρέπει να υπάρχουν τέτοιες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες. Αναφερθήκαμε επίσης και στη λήψη αποφάσεων και επίσης αναφερθήκαμε και στα παιδιά με αναπηρίες και τονίσαμε το ότι η εκπαίδευση ε, θα πρέπει να προσφέρεται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν πρόσβαση και τα παιδιά με αναπηρίες. Αναφερθήκαμε τέλος και στις δημόσιες συμβάσεις. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι με όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα, αγγίξαμε όλες τις πτυχές της ζωής. Πριν από ένα χρόνο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Απασχόληση και τις Κοινωνικές Υποθέσεις, εγκρίναμε ένα ψήφισμα για την κινητικότητα των ατόμων με αναπηρίες και, για την ένταξή τους ήταν το κείμενο αυτό. Σήμερα αναφερθήκαμε πολλές φορές στην κινητικότητα και γι' αυτό είμαι περήφανος που βοήθησα και εγώ στη σύνταξη της έκθεσης αυτής. Συνεργάστηκα βέβαια με άλλους 34 ευρωβουλευτές και μίλησα προηγουμένως με πάρα πολλούς εκπροσώπους οργανώσεων που ασχολούνται με τα θέματα των ατόμων με αναπηρίες. Πρέπει να φροντίσουμε στο μέλλον, ό,τι και αν κάνουμε, να έχουμε και τη συμμετοχή των ε, ατόμων με αναπηρίες. Τώρα προσβλέπουμε και στην ε, Ευρωπαϊκή Πράξη για την ε, Προσβασιμότητα και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία αναφέρθηκε στη σημασία που έχει η πράξη αυτή. Πριν από ένα χρόνο, πρέπει να σας πω, Ακούσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθούσε πρόταση για την πράξη αυτή προσβασιμότητας. Δυστυχώς όμως δεν έχει γίνει αυτό ακόμα. Ανταυτού πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε μία πράξη πάνω στο τραπέζι που να είναι όμως λεπτομερής. Να μην έχει ασαφείς νομικές προδιαγραφές. Και χαίρομαι που σήμερα εγκρίναμε το ψήφισμά μας. Δεν γνωρίζω επακριβώς το περιεχόμενο, αλλά είμαι σίγουρος ότι περιλαμβάνει πολύ σοβαρές προτάσεις. Και εμείς στη διακυκομματική ομάδα να ξέρετε ότι θα το συζητήσουμε και θα ανταλλάξουμε απόψεις μεταξύ ευρωβουλευτών. Και στη συνέχεια ελπίζουμε ότι θα ετοιμάσουμε και εμείς ένα ψήφισμα το οποίο θα πιέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να λάβουν υπόψη τους τα όσα ζητάνε τα άτομα με αναπηρίες και ότι θα γίνουν σωστές προτάσεις. Κατόπιν τούτων, ελπίζω να έχουμε μία απόφαση για τα επόμενα 7 χρόνια σχετικά με τα κονδύλια, έτσι ώστε να υπάρχουν αρκετά χρήματα. Αύριο και μεθαύριο θα γίνουν πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις. Ελπίζω ότι οι ευρωβουλευτές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις θα ε, αποφασιστικά θα υποστηρίξουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Θέλουμε να σας ενθαρρύνουμε γι' αυτό. Οι προτάσεις σας ε, πάντως είναι κάτι και θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και τώρα και στο μέλλον. Είναι κάτι αναγκαίο ζωτική σημασία για μας γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμα αυτό και πιο πέρα. Η ευρωπαϊκή πολιτική αλλιώς δεν θα έχει αξιοπιστία. Είναι τιμή για μένα που μπόρεσα σήμερα να συνεργαστώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ, Άνταμ. Ευχαριστώ όλους που βρεθήκατε εδώ σήμερα για το σημαντικό σας έργο. Συνεχίστε. Και θα σας διαβεβαιώσω ότι παρότι φεύγουμε από το Κοινοβούλιο, οι ιδέες σας, οι ιστορίες σας, τα αιτήματά σας θα παραμείνουν σε αυτό το Κοινοβούλιο. Θα ακολουθήσουμε τα βήματά σας μέσα στους επόμενους μήνες και τις επόμενες μέρες. Επίσης θα ήθελα να σας στείλω ένα μήνυμα σε όσους βρισκόνται επίσης στην του ευχαριστούμε και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο. Έτσι εδώ μου δόθηκε με μια ευκαιρία να κλείσω τη σύνοδο αυτή και θα σας αναφέρω τα λόγια του αγαπημένου μου ε, ποιητή. Τα λόγια του περσινού χρόνου ανήκουν στον περσινό χρόνο το να φτάνει κανείς ένα τέλος σημαίνει μια νέα αρχή. Αυτά είναι τα λόγια του T.S. Eliot και από μένα εδώ ολοκληρώνω τη συνεδρία σας. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα, καλή χρόνια και μια νέα καινούργια αρχή για το έργο σας για το επόμενο έτος. Εδώ δίνω τον λόγο στον κύριο Γιάννη Βαρδακαστάνη, ο οποίος επίσημα θα κλείσει τη σε αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν εντυπωσιακή η σημερινή ημέρα. Γεμάτη αποφασιστικότητα. Μια μέρα κατά την οποία στείλαμε ένα ισχυρό, καθαρό μήνυμα στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους ηγέτες των χωρών μας. Ότι εμείς, τα άτομα με αναπηρίες και οι οικογένειές μας δεν θα ανεχτούμε και δεν θα δεχθούμε να είμαστε τα πρώτα θύματα των μέτρων λιτότητας. Θεωρούμε τα μέτρα λιτότητας ως άμεσες παραβιάσεις και καταχρήσεις των δικαιωμάτων που θεσπίζονται στην Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες. Η σημερινή ημέρα είναι ιστορική.

να καταστήσει παράνομες τις διακρίσεις να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα που απαιτούνται για την προστασία, την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες. Σήμερα είναι πιο σημαντικό από ποτέ να υλοποιηθούν όλα αυτά, διότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια ταραγμένη εποχή, σε μια βαθιά οικονομική, κοινωνική κρίση που όπως είπατε πολλοί από εμάς, αν όχι όλοι μας βλέπουμε πλέον ως κρίση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πέρυσι, στις 6 Δεκεμβρίου έλαβε χώρα η πρώτη συνάντηση ε, ενημέρωσης για άτομα με αναπηρίες. Τα οι τρεις πρόεδροι των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων μαζί με το EDF ε, συζήτησαν το πώς η συνθήκη για τα άτομα με αναπηρίες των ΗΕ θα μπορούσε να υλοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία από τις δεσμεύσεις που έγιναν τότε ήταν ότι θα λάμβανε χώρα το Τρίτο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα άτομα με αναπηρίες. Αυτό που έλαβε χώρα σήμερα. Αλλά έγιναν και άλλες δεσμεύσεις. Δεσμεύσεις που θα χρειαστεί να εκπληρώσουν τα θεσμικά όργανα και οι ηγέτες των θεσμικών όργανων γνωρίζουν ότι ένα από τα χαρακτηριστικά του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τους αναπήρους είναι ότι δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε έτσι λοιπόν για το επόμενο έτος να το γνωρίζετε κι εσείς ε, και αυτά είναι συμπεράσματα από τα όσα συζητήσαμε το επόμενο έτος θα επιδιώξουμε μια συνάντηση όλων των επιτρόπων όπως μας υποσχέθηκε ο Πρόεδρος Μπαρόσο ώστε να συζητήσουμε την υλοποίηση τη συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης Επιδιώκουμε τη δεύτερη και ενημέρωση για τα άτομα με αναπηρίες για το επόμενο έτος, το State of the Union, διότι έγινε δέσμευση ώστε να λαμβάνει η χώρα αυτό το State of the Union κάθε δεύτερο έτος. Δηλαδή μέχρι το Δεκέμβριο του 2013 θα πρέπει να έχει λάβει η χώρα ξανά. Νωρίτερα σήμερα έκανα την πρόταση στον αρχηγό της ομάδας των σοσιαλιστών και στον αντιπρόεδρο του ΕΛΚ του Κοινοβουλίου να συναντηθούν παρουσία μας σε μια συνάντηση των ηγετών των πολιτικών ομάδων του Κοινοβουλίου ώστε να συζητήσουμε το ψήφισμα που εγκρίναμε σήμερα. Διότι άλλο ένα χαρακτηριστικό δικό μας είναι ότι μας αρέσουν τα ψηφίσματα αλλά δεν τα θεωρούμε δηλώσεις. Θεωρούμε τα ψηφίσματα ως δεσμεύσεις. Θέλουμε να υλοποιηθούν. Θέλουμε να τα υλοποιήσουν. Θέλουμε λοιπόν να συζητήσουμε με τους αρχηγούς των πολιτικών ομάδων το πώς τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες θα τεθούν πιο ψηλά στην ατζέντα όχι μόνο του Κοινοβουλίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των συνολό Σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες θα πρόκειται να συναυθούν του χρόνου διαρθρωτικά ταμεία, εξωτερική αρρωγή κτλ. κτλ. Αλλά και νέε. Η νομοθεσία για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο έχει ήδη δημοσιοποιηθεί η πρόταση. Αναμένουμε την Ευρωπαϊκή Πράξη Προσβασιμότητας και άλλες πρωτοβουλίες τις οποίες θα δούμε του χρόνου. Του χρόνου λοιπόν, το επόμενο έτος είναι ένα έτος όπου θα ξεκινήσουμε να υλοποιούμε το ψήφισμα το οποίο εγκρίναμε σήμερα. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους εργάστηκαν σκληρά ώστε η σημερινή ημέρα να γίνει πραγματικότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υποστήριξη που παρέχει το Κοινοβούλιο. Πολιτική, οικονομική, διοικητική υποστήριξη. Τον ευχαριστώ που μας έδωσε, μας παραχώρησε τους χώρους για τις συναντήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου, όλους τους ευρωβουλευτές που ήταν μαζί μας σήμερα, την πολύ ενεργό συμμετοχή των μελών οργανώσεων για άτομα με αναπηρίες και κυρίως τον πρόεδρο της διακομματικής ομάδας ε, Άνταμ Κόσε για άτομα με αναπηρίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη της γραμματείας του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για άτομα με αναπηρίες που εργάστηκαν αδιάκοπα για να γίνει η σύνοδος αυτή πραγματικότητα. Οι ευρωβουλευτές, ε, τα μέλη των εθνικών οργανισμών, τα μέλη του EDF που έφεραν εδώ τις αντιπροσωπείες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους Δερμινείς. Όχι μόνο επειδή βοήθησαν, μας βοήθησαν να επικοινωνήσουμε όλους τους Δερμινείς και της νοηματικής, αλλά και για την υπομονή τους. Την υπομονή που έδειξαν μαζί μας. Και θα ήθελα να ολοκληρώσω και εγώ με ένα ποίημα ένα απόσπασμα από ένα ποίημα το οποίο χρησιμοποιώ σε περιπτώσει σαν αυτήν. Υπάρχουν μερικοί που ζουν στο σκοτάδι, ενώ άλλοι ζουν στο φως. Βλέπουμε αυτούς στο φως της ημέρας, εκείνους. Στο σκοτάδι τους βλέπουμε εκτός. Είναι αόρατη, Μπέρτολτ Μπρέχτ. Είναι αποστολή. Είναι καθήκον του κινήματος για τα άτομα με αναπηρίες σε όλα τα επίπεδα να φέρουμε τους συναδέλφους μας στο φως μακριά από το σκοτάδι Έχουμε μια ασφαλή επιστροφή σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα χαρούμενο νέο έτος δραστήριο νέο έτος προενεργό νέο έτος και αν χρειαστεί κατεβείτε στους δρόμους καταστήστε σαφές ότι δεν είστε παθητικοί. Δεν είμαστε παθητικοί. Δεν είμαστε αποδέκτες εξυπηρετήσεων. Έχουμε δικαιώματα. Το μήνυμα είναι καθαρό. Το μήνυμα είναι ηχηρό. Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς. Ευχαριστώ.